Ladies and gentlemen, welcome. και κύριοι, καλώ ορίσατε. Παρακαλώ καθίστε. Ladies Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε σε αυτή την ακρόαση που φέρει τον τίτλο «Διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων, ρυθμιστικές πτυχές και ε, ρυθμίσεις περί διαφορών μεταξύ επενδυτή και κρατών καθώς και διατησία». Καλωσορίζω τους εκπροσώπους της Επιτροπής ε, Διεθνούς Εμπορίου που συνδιοργανώνουν μαζί μας αυτήν την ακρόαση, μαζί με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, της οποίας έχω εγώ την τιμή να προεδρεύω. Αυτή η ακρόαση ακολουθεί μια άλλη που είχε γίνει στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων τον περασμένο Φεβρουάριο με τίτλο ε, «Ρυθμιστική συνοχή και εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας στο πλαίσιο της συμφωνίας TTIP». Η εξέβρεση μιας γενική συμφωνίας ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Ένωση όσον αφορά τι ρυθμιστικέ επιτυχίε που περιλαμβάνονται στι διαπραγματεύσει της ΤΥΠΑ θεωρούνται σημαντικές, ουσιώδεις, στο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ε, στα μεμονωμένα τομεακά ζητήματα. Γι' αυτό και τα πάνελ θα έχουν δύο προσεγγίσεις στη σημερινή ακρόαση. Μία θα είναι ακαδημαϊκής φύσεως, όπου θα συζητάτε η πρόοδος των διαφόρων ε, τομέων από πλευράς ε, οριζόντιας και μια πρακτική προσέγγιση που από σημείο κίνηση θα είναι τα διάφορα πρακτικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες όσον αφορά τεχνολογία, τις παραγωγικές μεθόδους, την ασφάλεια καθώς και το περιβάλλον. Επιπλέον, της περαιτέρω συζήτηση των ρυθμιστικών πτυχών της ΔΥΤΥΠ, η σημερινή ακρόαση θα περιλαμβάνει και ένα πάνελ που θα εστιάσει στη νομική συζήτηση που αφορά τις πιθανές επιλογές για τη ρύθμιση διαφορών σύμφωνα με το διαθέσεις δίκαιο που ήδη υπάρχουν ή που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για τη TTIP και παρόμοιες συμφωνίες συμπεριλαμβανομένων των εθνικών δικαιοδοσιών, ρύθμιση διαφορών από κράτος σε κράτος, ρύθμιση διαφορών ανάμεσα σε επενδυτή και κράτος, ISDS σε διάκριση, σε αντίθεση με τα ισχύοντα υπό τις διμερείς συμφωνίες των κρατών μελών, καθώς και η διαβούλευση TTIP και πολιτών καθώς και η χρήση διεθνών οργανισμών όπως ο ΠΟΕ πιθανά ε, σε ε, πιθανά δικαστήρια διαθέσεις διεθνών διαφορών, διαμεσολαβήσεις κτλ. Η Επιτροπή ΙΝΤΑ είναι υπεύθυνη στο Ευρωκοινοβούλιο για τα ζητήματα που αφορούν εμπορικές συμφωνίες που διέπουν οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες καθώς και με περιφερειακούς οργανισμούς ενώ η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων είναι υπεύθυνη για την ερμηνεία, εφαρμογή και παρακολούθηση της κοινοτικής νομοθεσίας και της συμμόρφωσης με την κοινοτική νομοθεσία, ερμηνεία και εφαρμογή διεθνούς νομοθεσίας όσον αφορά την ε, επίδραση στην Ευρωπαϊκή Ένωση από καλύτερη ε, νομοθεσία καθώς και μέθοδοι ρύθμισης ε, ε, πολιτικών υποθέσεων, αστικών μάλλον υποθέσεων. Κοινή λοιπόν ακρόαση για να μπορέσουμε να έχουμε την εμπειρογνωμοσύνη ε, των ε, βουλευτών αλλά και του υποστηρικτικού προσωπικού των δύο επιτροπών. Στον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων TTIP που θα γίνει στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα θα μπορούμε να εστιάσουμε στις, ε, στα θέματα ε, σύγκρισης μεταξύ των διαφόρων νομοθεσιών. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στον Μπέρντ Λάγκε για τις εισαγωγικέ του παρατηρήσεις και έτσι ώστε να προεδρεύσει στο πρώτο πάνελ το οποίο θα αφιερωθεί στην ε, διαιτησία και ISDS. Ευχαριστώ Ταμάλα. Αγαπητέ κύριε Σφόμποτα, σας ευχαριστώ Ευχαριστώ και τους αγαπητούς συναδέλφους. Είναι μια πολύ καλή πρακτική να μπορούμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε τα θέματα τα οποία μας αφορούν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι σημαντικό να υπάρξει και σε νομικό επίπεδο ε, κάποια σύνδεση και κάποια συνάφεια με το δίκαιο το οποίο θέλουμε να εξασφαλίσουμε στη Συμφωνία TTIP Έχουμε δύο σημεία τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Καταρχήν το θέμα των δυνατοτήτων προστασία των ε, επενδυτών μέσω του ISDS, δηλαδή τη διαρρύθμιση διαμαχών μεταξύ επενδυτών και κρατών και επίση η συνεργασία σε ρυθμιστικό επίπεδο. Αυτά τα δύο θέματα τα οποία μα απασχολούν κυρίω. Στην επόμενη εβδομάδα θα λάβει χώρα 8 γύρο διαπραγματεύσεων όπου θα τεθεί ιδίω το θέμα τη ε, συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών και επίσης έχουμε τα πορίσματα της ε, διαβούλευσης που οργάνωσε η Κομισιόν και επομένως είμαστε υποχρεωμένοι να αντλήσουμε και τα πολιτικά συμπεράσματα από αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης. Τρίτον, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρουσιάσουμε μια ενδιάμεση έκθεση, ένα ενδιάμεσο ε, κατά κάποιο τρόπο ισολογισμό σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις της TTIP, όπου όλες οι εμπλεκόμενες επιτροπές θα πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία που άπτονται της δικής τους εμπειρογνωμοσύνης. Είναι υπό επεξεργασία αυτό, αυτό το ψήφισμα και θα έρθει στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Μάιο. Και έρχομαι τώρα στο πρώτο σημείο της ακρόασής μας, που είναι ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο στην συζήτηση που λαμβάνει η χώρα στην κοινή γνώμη, που είναι οι δυνατότητε προστασία των επενδυτών. Όπω ανέφερε ο κ. Σβόμποντα, δεν πρόκειται μονάχα για το θέμα τη διαιτησία μεταξύ κρατών και επενδυτών, αλλά τίθεται γενικότερα το ζήτημα του πώ θα μπορέσουμε να αρθρώσουμε μια λογική νομοθεσία η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία των επενδυτών και πιστεύω ότι υπάρχει μια ευρύτατη συνένεση μεταξύ όλων αυτών οι οποίοι έχουν λάβει, χώρα, έχουν λάβει μέρος μάλλον στην συζήτηση ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε με την εμπορική αυτή συμφωνία ότι θα υπάρχει προστασία των επενδυτών και όχι διάκριση εναντίον τους. Αυτό αφορά τους Ευρωπαίους στο εξωτερικό αλλά και τους επενδυτές από έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν επενδύουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2009 μέσα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρμοδιότητα, συναρμοδιότητα για συνθήκες αυτού του είδους λόγω της Ειδικής Λισαβόνας και το συμπέρασμα είναι ότι εμείς θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα κατάλληλα μέσα και οι κατάλληλες επιλογές τις οποίες θα πρέπει να καταλήξουμε μέσα στη συμφωνία αυτή. Έχουμε ήδη τις ε, συμφωνίες με τον Καναδά, υποδιαπραγμάτευση με την Σιγκαπούρη και τώρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες τίθεται το θέμα αυτό της προστασία των επενδυτών και έχουμε και συμφωνίες με την Μιανμάρ ε, και την Κίνα μόνο για θέματα επενδυτών και επίσης υπάρχει και μια συμφωνία με την Νότια Κορέα που έχει και αυτή ε, επιπτώσεις για τα θέματα των επενδυτών. Υπάρχουν λοιπόν οι ανάγκες να έχουμε μια συμβατή συμβατική ομοιομορφία στα θέματα αυτά και επίσης ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτή τη στιγμή ενώπιόν της περίπου 400 συμφωνίες ε, του είδους αυτού του επενδυτικού από το 2009. Έχουμε την νομοθεσία από το 2012 στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μας υποχρεώνει όλες αυτές οι 1.400 συγγνώμη συμφωνίες να ελεγχθούν κατά πόσο είναι σύμμορφες με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λοιπόν καταδεικνύουν τον κεντρικό χαρακτήρα αυτού του ζητήματος για την ευρωπαϊκή πολιτική και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε σήμερα μαζί μας τέσσερις εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα διαλάβουν ιδιαίτερα το θέμα της προστασίας των υπεδητών, ποια είναι τα καλύτερα μέσα για την προστασία των υπεδητών. Επομένως, δεν είναι μονάχα το θέμα της ε, ISDS, της ε, προστασίας της ε, επίλυσης διαφορών υπεδητών κράτους, αλλά θα είναι ε, γενικότερο το θέμα και θέλω να ξεκινήσω με τον εμπειρογνώμονα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο ε, Σλέγγελμιλ. Σας ευχαριστώ πολύ και σύμφωνα μαζί σας κύριε Λάγκε ότι η συζήτηση σε σχέση με λογικά επίπεδα προστασίας των επενδυτών τα οποία θα πρέπει να συνάδουν με τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει. Έχουμε δει ότι έγινε ήδη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγώ είμαι έτοιμος να επανέλθω στα βασικά προβλήματα αυτού του θέματος και να παρουσιάσω τη δική μας εικόνα σε σχέση με το ISDS και γενικότερα τα θέματα προστασίας των επενδυτών. Τι είναι το ISDS καταρχήν. Το πρώτο πράγμα το οποίο θέλω να αναφέρω. Δεύτερον θέλω να έρθω στο ζήτημα του γιατί προστατεύουμε τους επενδυτέ. Ένα τρίτο στοιχείο θα είναι κάποιε βασικές αρχές σε σχέση, βασικά στοιχεία για το ISDS. Και έρχομαι στα επιχειρήματα υπέρ και κατά σε σχέση με το ISDS. Και τέλος θα καταλήξω στο συμπέρασμα ότι για την Κομισιόν αυτή τη στιγμή η λύση πρέπει να είναι μεταρρύθμιση του συστήματος ISDS και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Καταρχήν, τι είναι το ISDS. Νομίζω ότι είναι μια απλή ερώτηση που μπορεί να ετύχει απλής απάντησης. Είναι ένας μηχανισμός για να υλοποιούνται ορισμένες διεθνούς χαρακτήρα υποχρεώσεις. Πρόκειται για ένα στενό τμήμα υποχρεώσεων που είναι καταρχήν η υποχρέωση να μην υπάρχουν διακρίσεις έναντι επενδυτών οι οποίοι έχουν επενδύσει στο έδαφος ενός κράτους. Δεύτερον, να μην υπάρξει ε, απαλωτρίωση των επενδύσεών τους χωρίς σωστή αποζημίωση και χωρίς κοινοφελή λόγο. Τρίτον, να μην υπάρχει ε, αρνησιδικία σε σχέση με τους επενδυτές και τέταρτον να υπάρχει η δυνατότητα εισόδου και εξόδου κεφαλαίων απροσκόπτως από τη χώρα επενδύσεων. Όλα αυτά λοιπόν θέλω να τα τονίσω ότι το καθεστώς των επενδυτών έχει ξεχωριστά χαρακτήρα. Ε, αυτές οι ρυθμίσεις δεν αφορούν άλλες υποχρεώσεις βάσει της συνθήκης εμπορίου, δεν έχουν να κάνουν με θέματα παραγωγικά δημοσίων ε, προμηθειών, ούτε για θέματα ε, συνεργασίας δημιουργικών αρχών που θα επανέλθουμε σε αυτά στη συνέχεια. Μόνο στην περίπτωση του ISDS είναι εφαρμόσιμες τέτοιες ρήτρε. Και δεν πρόκειται για αποζημίωση, για κέρδη που δεν πραγματοποιήθηκαν. Η προστασία από την απαλωτρίωση είναι ένα πράγμα, αλλά δεν μπορεί κανεί να προστατεύσει ένα παιδιτή για αλλαγή του επιχειρηματικού κλίματο. Δεύτερο ερώτημα, γιατί υπάρχουν τώρα όλοι αυτοί οι κανόνε. Για μένα, η κύρια διαφορά εναντί άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων είναι το γεγονός ότι οι επενδύσεις είναι δέσμευση μακροχρόνια. Μπορείτε να στείλετε τα εμπορευματοκιβώτια σας κάπου αλλού αν υπάρξει ένα εμπορικό πρόβλημα. Δεν μπορείτε όμως να μετακομίσετε το σύνολο των επενδύσεών σας, αν έχετε κάνει μια αγιώτηση δεν μπορείτε να τη μεταφέρετε κάπου αλλού ή αν έχετε επενδύσει σε ένα δίκτυο τηλεπικοινωνιών δεν μπορείτε την υποδομή να την πάτε κάπου αλλού. <clears throat> Είναι λοιπόν η επένδυση μια μακροχρόνια δέσμευση σε μια τρίτη χώρα και έχει διαφορετικό χαρακτήρα από μια εμπορική συναλλαγή και εάν υπάρχει κατάλληλη προστασία αυτό φυσικά κάνει πιο ελκυστικό ένα χώρο επενδύσεων αν υπάρχουν ορισμένες προδιαγραφές και ορισμένα είδη προστασίας προτού γίνει η επένδυση στο χώρο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Αναφέρατε κύριε Λάγκε ότι τα κράτη-μέλη μας έχουν ε, εγκρίνει περίπου τις μισές συμφωνίες αυτού του είδους στον κόσμο, από τις 3.000 αυτές συμφωνίες, 1.400, και αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους μεγαλύτερους επενδυτές σε παγκόσμιο επίπεδο, ε, εμείς και μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως, είμαστε και ο κύριος χρήστης αυτού του συστήματος. Οι πάνω από μισές από τις περιπτώσεις, τις νέες περιπτώσεις που είχαν, είχαν λάβει χώρα το 2014 αφορούσαν ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, κυρίως η περίπτωση της Repsol στην Αργεντινή, της πετρελαϊκής αυτής εταιρείας. Εκεί λοιπόν βλέπουμε γιατί υπάρχει ενδιαφέρον για περιπτώσεις που εμπλέκουν ευρωπαϊκές εταιρείες. Αν δούμε τώρα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα στην πράξη και το ερώτημα του κατά πόσο τίθεται σε κίνδυνο η κυριαρχικότητά μας σε επίπεδο ρύθμισης, και μαζί μου έχω τον ερευνητή ο οποίος έχει ασχοληθεί σε μεγάλο βαθμό για τα θέματα αυτά, 90% των περιπτώσεων δεν αφορούν νομικές υποθέσεις. Είναι προσφυγές εναντίον διοικητικών μέτρων εφαρμογής της νομοθεσίας. Οι τοπικές αρχές μπορούν να πάρουν μια απόφαση, μια περιφέρεια μπορεί να άρει μια αδειοδότηση και οι υπόλοιπες 10% δεν αφορούν όλες θέματα νομοθεσίας και εξάλλου δεν είναι μονάχα οι μεγάλες πολυεθνικές οι οποίες εμπλέκονται σε τέτοιες διαδικασίες. Φαίνεται ότι 45% των μεσαίων εταιριών ε, εμπλέκονται και 22% είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχετε ακόμα και περιπτώσεις που ένας ιδιώτης μπορεί να προσφύγει εναντίον ενός κράτους. Ας έρθουμε τώρα στα κύρια επιχειρήματα υπέρ του τρόπου αυτού παροχής ε, θεραπείας και προστασίας τους επενδυτές. Καταρχήν, ε, το βασικό μας επιχείρημα είναι ότι πρέπει να γίνονται οι επιλύσεις των προβλημάτων αυτών από τα εγχώρια δικαστήρια. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι διεθνείς υποχρεώσεις προστασίας των επενδυτών δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμες σε τοπικά δικαστήρια δεν υπάρχει το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των ρητρών και υπάρχει ένας απλός λόγος γι' αυτό. Τα εθνικά δικαστήρια δεν θέλουν να εφαρμόσουν το διεθνές δίκαιο και τα εγχώρια δικαστήρια μπορούν να ακυρώσουν ένα μέτρο διεθνούς χαρακτήρα και δεν θέλει κανείς να γίνεται κάτι τέτοιο. Το ISDS αφορά μονάχα τα θέματα της αποζημίωσης για τα εγχώρια δικαστήρια και επίσης οι ΗΠΑ έχει αρνηθεί το άμεσο αποτέλεσμα και επειδή δεν υπάρχει αμοιβαιότητα με άλλες χώρες, ούτε και εμείς θέλουμε να ισχύει κάτι τέτοιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο θέμα, και εδώ επαναλαμβάνω εν μέρει αυτό το οποίο είπα προηγουμένως, είναι το εξή Όταν μία διεθνής υποχρέωση δεν έχει άμεσο αποτέλεσμα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, Δεν μας βοηθάει η ευρωστία του τοπικού δικαστικού συστήματος. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι καλά τα τοπικά δικαστήρια θα λύσουν το πρόβλημα γιατί εφαρμόζουν μονάχα το τοπικό, το εγχώριο δίκαιο και όχι το διεθνές. Στις ΗΠΑ δεν υπάρχει καμία απαγόρευση για διακρίσεις. Βλέπετε ότι οι νόμοι περί προμηθειών και άλλοι νόμοι εφαρμόζουν διακρίσεις θετικές περί των ΗΠΑ. Επομένως δεν μπορούμε να ελπίζουμε να υπάρχει μια τέτοια ρήτρα σε μια εμπορική συμφωνία. Ένα άλλο παράδειγμα, επειδή μιλάμε και για τη συμφωνία TTIP, οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν καταθέσει περισσότερες προσφυγές κατά του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, 130 περίπου, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, για θέματα αυτού του είδους. Και θεωρούν ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το τοπικό ε, σύστημα το δικαστικό ένα τέτοιο, τα προβλήματα αυτού του είδους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντίθετα έχει ένα ισχυρό σύστημα προστασία και μα ενδιαφέρει αν δεν υπάρχει δυνατότητα προσφύγή σε εθνικό δικαστήριο να υπάρχει και μία άλλη δυνατότητα προσφυγή. Ένα άλλο επιχείρημα που αναφέρεται είναι γιατί δεν χρησιμοποιείται συστήματα επίλυση διακρατικών διαφορών. Γιατί πρόκειται εδώ για συνθήκε ε, από τις οποίες απορρέουν οι υποχρεώσεις. Αλλά 90% των περιπτώσεων έχουν να κάνουν με διοικητικά μέτρα. Αν χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία επίλυση διαφορών στον ΠΟΕ μεταξύ κρατών, αυτό αφορά μόνο λίγες περιπτώσεις και είναι συστημικές περιπτώσεις που έχουν σημαντικό εμπορικό αντίκτυπο. Δηλαδή σε επίπεδο διακρατικό δεν θα μπορούσαμε να διεκπαιρεώσουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις γιατί δεν έχουν συστημικό ε, ενδιαφέρον. Μιλάμε για μεμονωμένες εταιρείε συνήθως. Και επίσης δεν είναι ελκυστικό αυτό το σύστημα για τους επενδυτές μας γιατί θα πρέπει να διαλέξουμε ποιες περιπτώσεις θα φέρουμε στον ΠΟΕ θα πρέπει να υπάρξει και διευθυνσία για τα κράτη-μέλη μεταξύ των κρατών μιλών για τα θέματα αυτά και όλα εξαρτώνται από την καλή θέληση των κυβερνήσεων να λύσουν μια διαφορά η οποία είναι ουσιαστικά μια διαφορά μεταξύ εταιριών στην πράξη. Θα κάνει πιο δύσκολο αυτό για μικρές χώρες να μπορέσουν να φέρουν στην προσοχή των κυβερνήσεών τους ή στην προσοχή του ΠΟΕ τα θέματα αυτά και κινδυνεύει να υπάρξει έλλειψη προστασίας. Το γεγονός λοιπόν ότι το βασικό μοντέλο του ISDS ότι δηλαδή ο ίδιος ο επενδυτής μπορεί να κάνει μια προσφυγή εναντίον ενός κράτους είναι η καλύτερη λύση για το συγκεκριμένο αυτό τομέα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το σύστημα το ίδιο είναι τέλειο, κάθε άλλο. Έχουμε προφανώς εντοπίσει μια σειρά από προβλήματα όπου περιπτώσει όπου θεωρούμε ότι το σύστημα μπορεί να βελτιωθεί και το έχουμε τονίσει και σε συζητήσεις εναντίον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι το σχέδιο συμφωνία μα με τον Καναδά και τη Σιγκαπούρη μας δίνουν ένα τέτοιο παράδειγμα. Δίνουν πλήρη διαφάνεια για να αντιμετωπίσω μια επίκριση. Είναι αποτελεσματικά συστήματα γιατί υπάρχουν ανεξάρτητοι διαιτητές και εξασφαλίζουν και αποτελεσματική εποπτεία από τα κράτη-μέλη. Θα σας δείξω στο τέλος και μια διαφάνεια για αυτούς που ενδιαφέρονται για τις λεπτομέρειες έχει ορισμένε στήλε που δείχνει όλες τις βελτιώσεις που έχουμε επιφέρει ε, στο αρχικό σχέδιο της συμφωνίας μετά την σύναψη της συμφωνίας της ε, Λισαβόνας. Έχουμε και την ε, διαβούλευση η οποία έλαβε χώρα, όπως αναφέρθηκε από τους Πρόεδρους. Κάναμε μια διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών και τους εμπλεκομένους ήταν μάλλον σκεπτικιστική η αντίδραση των περισσότερων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση, αν δεν ήταν συντριπτικά σκεπτικιστική, αλλά συγχρόνως πολλοί έχουν παράσχει σημαντικά, σημαντικές ιδέες για βελτίωση του συστήματος και έχουμε τέσσερις τομείς όπου θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο στο μέλλον. Κατά την απόψή μας η μεταρρύθμιση θα πρέπει να εστιάσει σε μια καλύτερη προστασία του δικαιώματος ρύθμισης. Δεύτερον, να μπορέσουμε να δούμε την ε, εδραίωση και τη λειτουργία των ε, διαιτητικών δικαστηρίων, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή, τρίτον, θα πρέπει να δούμε πιο προσεκτικά πώς τα εθνικά ε, δικαστικά συστήματα θα μπορέσουν να αλληλεπιδρούν για να μην υπάρχουν παράλληλες προσφυγές και να υπάρχει μια σαφέστερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ τους και τέταρτον νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη συνένεση ότι χρειάζεται ένα εφετείο κατά κάποιο τρόπο, ένα δεύτερο σώμα προσφυγής, ένα δευτεροβάθμιο σώμα προσφυγής μετά από το πρωτοβάθμιο διαιτητικό δικαστήριο. Όλα αυτά θέλω να σας πω και ευχαριστώ για την προσοχή σας. That, that was σας ευχαριστώ, ήταν ξεκάθαρα τα όσα είπατε. Άρα, η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολουθεί η κυρία Φρέια Μπέτενς, που είναι καθηγήτρια δικαίου στο Πανεπιστήμιο Λέιντεν και είναι και δικηγόρος στο δικηγορικό σύλλογο. Έχει το λόγο κυρία μου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου πρώτα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω και τις θεωρητικές πτυχές, γιατί με τα πρακτικά που ανέπτυξε προηγουμένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνώ. Με συγχωρείτε. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω τρία πράγματα. Πρώτο, ποιο είναι ο λόγο που έχουμε την ISDS και νόμους για προστασία των επενδύσεων. και κάποιες παρανοήσεις που επανέχονται σε εκθέσεις και στη συζήτηση αυτή. Και αν εξετάσετε το κόστος και όφελος, Να ποια ωφέλη μπορούν να υπερβαίνουν ποια, ε, ποιο κόστος. Και πρώτα, γιατί χρειαζόμαστε το σύστημα αυτό. Δημιουργήθηκε το σύστημα αυτό ως αντίδραση κατά αυθαίρετων απαλωτριώσεων με την ιδέα να υπάρχει μια νομοθεσία που να προβλέπει τα ελάχιστα δικαιώματα των επενδυτών και να έχει παγκόσμια ισχύ. Γιατί δημιουργήθηκε η STS. Υπήρχε κατά κάποιο τρόπο μια διπλωματική προστασία γιατί σας παρήχε προστασία η χώρα σας. Αλλά αυτό τελικά ήταν αυθαίρετο, ήταν πολιτικού χαρακτήρα και τελικά ως ιδιώτης χάνατε πια το δικαίωμα στην ίδια σας την προσφυγή. Ποιες είναι οι επιλογές που προτάθηκαν. Αφενός να επανέλθουν σε ένα σύστημα διακρατικών διαιτησιών, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να επιτύχει, γιατί υπάρχει και έντονη οικονομική πτυχή και δεν θα έπρεπε να εντάσσεται εκεί, καθώς και η απόφαση μιας χώρας να υιοθετήσει την προσφυγή που δεν έχει τόσο σχέση με το αν έχει υποστεί βλάβη ο, επενδυτή, ο επενδυτής ή περισσότερο αν είναι σκόπιμο να επιτεθεί κατά της άλλης χώρας. Ορισμένες από τις κοινέ παρανοήσεις τώρα έχουν ως εξής το σύστημα αυτό δεν είναι για τη χρήση μόνο μεγάλων επιχειρήσεων, που χρησιμοποιούν πολύ και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι περισσότερες υποθέσεις κερδίζονται από το κράτος. Και όπου δεν κερδίζει ε, τελικά το κράτο, αλλά κερδίζει ο επενδυτής, οι αποζημιώσει είναι μικρότερες από αυτές που ήλπιζε ο ίδιο ο επενδυτής ή η επενδύτρια. Και οι περισσότερε υποθέσει έχουν κινηθεί από επενδυτέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως από την Ολλανδία, το Ενωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Και λιγότερες υποθέσεις, λιγότερες προσφυγές από Αμερικανούς. Και καμία προσφυγή δεν είχε γίνει εκτός από την υπόθεση Vattenfall που κατέληξε στις εφημερίδες γιατί ήταν πραγματικά η μεγάλη εξαίρεση. Όπως είπα πριν δεν πρόκειται τόσο για θέματα νομοθεσίας αλλά για αποφάσεις διοικητικές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και κατά αυτόν στρέφονται συνήθως οι πρόσφυγες. Όσον αφορά τώρα την ανάλυση κόστους κόστους-οφέλους, τα εθνικά μας δικαστήρια θα μπορούσαν να είναι επαρκή, λέγεται συχνά. Βέβαια υπάρχουν νόμοι και στις ΗΠΑ και στις χώρες της Ένωσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η προστασία που παρέχουν εφαρμόζεται, πάντα, εφαρμόζεται πάντα, γιατί συχνά υπάρχουν και πολιτικές ευαισθησίες και Καμιά φορά οι δικαστές και ιδιαίτερα οι ένορκοι έχουν μια πίστη προς ε, το κράτος, την πατρίδα τους δηλαδή, που υπαγορεύει κάπως ε, τις ε, αποφάσεις που λαμβάνουν. Και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε δει ότι τα εθνικά μας δικαστήρια δεν εφαρμόζουν πάντοτε το διεθνές δίκαιο. Πρόσφατα, μία μη κρατική οργάνωση προσπάθησε να προσφύγει ενώπιον του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά μια διεθνού συμφωνία και δεν έγινε δεχτή η προσφύγη αυτή. Αυτό δεν σημαίνει λοιπόν ότι τα δικαστηριά μα θα εφαρμόσουν πράγματι το διεθνέ δίκαιο. Συχνά επίση ένα επιχείρημα που ακούγεται είναι ότι αν έχουμε ένα καλό σύστημα, τι μα χρειάζεται τότε, αν έχουμε καλό εθνικό σύστημα δηλαδή, τι μα χρειάζεται το διεθνέ. Εγώ τότε ρωτώ, αυτό σημαίνει ότι αν θέλετε, για παράδειγμα, να καταργήσετε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επειδή όλε οι χώρε μέλη έχουν επαρκή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι λοιπόν θα το καταργήσετε τότε και τότε βέβαια αλλάζουν πολύ συχνά γνώμη οι συνομιλητέ μου. Η ιδέα τώρα για την ISTS ότι θα αναφέρεται στις πιο ξεκάθαρες υποθέσεις, θα εφαρμόζει πιο ξεκάθαρες υποθέσεις όπου δεν έχουν διορθώσει την κατάσταση χώρες μελή. Συχνά δεν είναι δυνατό αυτό να γίνει στο εθνικό επίπεδο και είναι πάλι μια συνήθις παρανόηση ότι οι εθνικές Δικαστικέ διαδικασίε είναι και φθηνότερε ή λιγότερο δαπανηρέ. Μην δυσμονείτε ωστόσο ότι στι περιπτώσει αυτέ το κράτος αναλαμβάνει να πληρώσει τα δικά του δικαστικά έξοδα. Όχι μόνο αυτά, αλλά και τα διαδικαστικά έξοδα. Και αν έχετε και πρώτο βαθμό, μετά έφεση σε δεύτερο βαθμό και ούτε καθεξή, μπορεί τελικά η υπόθεση να αποβεί πάρα πολύ δαπανηρή. Αυτό το επιχείρημα που προβάλλουν ορισμένοι λοιπόν μπορεί να ε, αντισταθεί πολύ εύκολα. Είναι λοιπόν καλό το σύστημα. Όχι. Υπάρχει χώρος για βελτίωση. Και μία από τις πιθανές βελτιώσεις είναι να διατυπωθεί η συνθήκη με τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει περιοριστική, περιοριστικό ορισμό του επενδυτή και των επενδύσεων. Δεν θέλετε να προστατεύσετε, για παράδειγμα, ε, εταιρείε ψευδεπίγραφης που έχουν μοναχά κάπου ένα ε, γραμματοκιβώτιο. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, την, ε, το τραπεζικό κλάδο που δεν εμπίπτει στην ε, συνθήκη αυτή. Η δίκαιη και η ισότιμη μεταχείριση είναι ωστόσο ως όρος αρκετά ε, ασαφής. Τι σημαίνει η ισοδίκαιη. Μπορούν να αποκλειστούν και ορισμένες προστασίες, για παράδειγμα τα δικαιώματα πρόσβασης στην αγορά. Τέτοιου είδους συνθήκες λοιπόν εφαρμόζονται και προστατεύουν επενδύσεις που ήδη υπάρχουν. Μπορούν να αποκλειστούν επίσης αυτές οι συνολικές ρήτρες, umbrella clauses, που συναποτελούν μέρος μιας, διεθνής, μιας διεθνούς συνθήκης όπου δεν αρμόζουν. Και σε ορισμένες αμερικανικές συνθήκες μπορεί να περιλάβει κανείς μια ρήτρα δημόσιας προστασίας. Για παράδειγμα, για προστασία τη υγεία του περιβάλλοντος, των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτό είναι δυνατό. Οι περισσότερες χώρες μέλη στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το έχουν πράξει ω τώρα. Πέρα από αυτό, είναι δυνατό να διαμορφωθεί έτσι η διαδικαστική πρόσβαση ώστε ο καθένα να έχει πρόσβαση στο σύστημα ISTS. Μια άλλη πρόταση θα ήταν να εξαντλούνται πρώτα τα τοπική, τοπική βαθμή δικαιοδοσία η εθνική βαθμή δικαιοδοσία πριν να φτάσει κανεί στη διεθνή διαιτησία. Αυτό είναι μια επιλογή. Θα μείωνε το ποσό των προσφυγών, μπορεί όμω να αυξήσει το κόστο του. Το κόστο του, γιατί θα πρέπει πρώτα να περάσουν από τι εθνικέ διαδικασίε και μετά καπέλο να έρθει και η διεθνή διαδικασία. Η διεθνή διαιτησία δηλαδή. Αν σκεφτείτε και πάλι το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μπορεί να περάσουν και 10 και 15 χρόνια από τον πρώτο βαθμό έχει τον τελευταίο. Μια άλλη επιλογή θα μπορούσε να είναι του σταυροδρομιού, δηλαδή ο επενδυτή δεν είναι υποχρεωμένο να επιλέξει είτε την εθνική διαδικασία είτε τη διεθνή διαδικασία, όχι και τα δύο. Άλλος τρόπος μείωσης των προσφυγών είναι η ε, ρήτρα προστασία απέναντι σε καταχρηστικές προσφυγές που να επιτρέπει να ε, απορρίπτονται εξ αρχής προφανώς αβάσιμες προσφυγές και να μην περάσουν από όλη την διαδικασία. Και αυτό βέβαια να συνδεθεί και με την αρχή the loser pays. Αυτός που χάνει τη δίκη δηλαδή αναλαμβάνει να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα. Ο επενδυτής εν τέλει δηλαδή εφόσον χάσει την δίκη να αναλάβει να πληρώσει και τα δικαστικά έξοδα του κράτους κατά του που προσέφυγε ή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άλλο που θα μπορούσε να ε, ε, προβλεφθεί θα είναι η διαμεσολάβηση η διαμεσολάβηση να είναι υποχρεωτική, να είναι πρόδρομος απέναντι στην ISDS, να μην αρχίζει δηλαδή να λειτουργεί η ISDS πριν να περάσει η φάση της διαμεσολάβησης. Άλλο στοιχείο του κόστους, της ανάλυσης κόστους είναι να μπουν κάποια προστατευτικά μέτρα μέσα στο ίδιο το σύστημα. Δηλαδή, να μη σημαίνει ότι τα κράτη ή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούν να αυτοπροστατευτούν. Και άλλος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να αυξηθεί η διαφάνεια. Για την ώρα οι ιδιωτησίες ανατίθενται και ιδιωτικά, αλλά να έχει κανείς πληροφορίες από πριν για τις ε, υποθέσεις, για τις διαφορές, για τους ισχυρισμούς που υποβάλλουν οι επενδυτές, ώστε να μπορεί ο κόσμος να παρακολουθεί τις υποθέσεις αυτές και τι ακριβώς γίνεται. Για παράδειγμα, στην συμφωνία ναύτα της Βόρειας Αμερικής, Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά, υπάρχει αυτό. Και πάει ο κόσμο και παρακολουθεί τι δίκε αυτέ. και εκεί πραγματικά οι πληροφορίε που λαμβάνει το κοινό είναι πολύ καλύτερη ποιότητας. Μα μπορείτε να μου πείτε ότι υπάρχουν κάποιε πληροφορίε που δεν θα θέλουμε να διαθέσουμε στο κοινό. Για παράδειγμα, για διαβαθμισμένε πληροφορίε κρατών ή και επιχειρήσεων και για του επενδυτέ. Αυτό όμως δεν κρίνεται από μόνο του, θα πρέπει να το κρίνουν τα δικαστήρια και να το εφαρμόζουν με τρόπο περιοριστικό. Άλλο, άλλη δυνατότητα είναι να έχουν ένα ενεργό ρόλο ε, κράτη-μέλη που είναι μέρη της, ε, της ε, συνθήκης, όχι όμως της διαφοράς. Το ίδιο για μη κρατικές οργανώσεις ή και για διεθνείς οργανώσεις ή άλλα, άλλες χώρες μέλη της Ένωσης. Επίσης μπορείτε να συμφωνήσετε ένα κώδικα δεοντολογίας. Ένα από τα παράπονα που ακούω για την ε, ISTS είναι ότι ένας μικρός αριθμός διαιτητών ε, κρίνει όλες τις υποθέσεις. Αυτό συμβαίνει διότι οι επενδυτές ορίζουν ξανά και ξανά τα ίδια πρόσωπα. Δεν είναι υποχρεωμένοι, αλλά αυτό κάνουν τελικά. Να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες για τις δημοσιοποιήσεις. Και επίση μπορείτε να συμφωνήσετε και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει τη σχετική πρόταση να υπάρχει ένα κατάλογος διαιτητών που να είναι συμφωνημένο από πριν, πριν να προκύψει η διαφορά, ότι αυτοί οι 30-40 άνθρωποι είναι καλοί διαιτητέ. Και αν θέλετε να διορίσετε κάποιον διαιτητή, θα πρέπει να πάρετε κάποιον ή κάποιον από αυτή τη λίστα. Επίσης, ένας μηχανισμός που θα προβλέπει, θα ενισχύσει την νομιμοποίηση και την προβλεψιμότητα του συστήματος και να προ, προλαβαίνει σφάλματα κακής εφαρμογής του νόμου. Δεν σημαίνει όμως ότι όλα τα κράτη, όλα τα μέρη ή κράτη ή και ε, επενδυτές θα προσφεύγουν ο Παγκόσμιο Οργανισμός Εμπορίου έχει όργανο προσφυγής, όπου προσφεύγουν δηλαδή αυτοί που χάνουν σε πρώτο βαθμό. Και υπάρχει και στην νομολογία και μπορεί να γνωρίζει κάποιο την αναμένη αναμένει σε περίπτωση που προσφύγει. Διαρκή δικαστήρια Καμιά φορά λένε ορισμένοι δεν θέλουμε διαιτητέ. μπορεί να θέλουμε ένα διαρκέ δικαστήριο. Αυτό είναι μια δυνατότητα. Υπάρχει ένα αριθμό τέτοιων διαρκών δικαστηρίων, μπορείτε να προσθέσετε κάτι τέτοιο στην ε, συνθήκη. Το ερώτημα είναι, το θέλετε πραγματικά αυτό, διότι σε αυτό το permanent court χρειαζόσατε και κτίριο, ε, γραμματική υποστήριξη, διαρκείς δικαστές. Αυτό βέβαια προσθέτει στις δαπάνες, χωρίς να προσθέτει απαραίτητα στην ποιότητα. Είναι μια επιλογή όμως. Τώρα, αν θα είναι ένα τέτοιο διαρκές δικαστήριο ανασύνθηκη, ανασύμβαση, αυτό πάλι δεν είναι απαραίτητο. Δεν θα είναι μονάχα, δεν θα πρέπει να συμφωνήσουν μονάχα οι Ηνωμένε Πολιτείε και η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να συμφωνήσουν και τα άλλα συμβαλόμενα μερική σου πολιτικά αυτό να μην είναι ρεαλιστικό. Έγινε προσπάθεια, για παράδειγμα, με πολυμερείς συμφωνίες ή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και φαίνεται ότι είναι ένα θέμα όπου δεν ε, υπάρχει πολυμερής ε, συνένεση. Αν λοιπόν ε, εξετάσετε αυτή την ανάλυση κόστους οφέλους, βλέπετε ότι πρώτα χρειάζεστε καλύτερες και πιο εκτεταμένες συνθήκες, συμβάσεις δηλαδή, που να ξεκαθαρίζουν απολύτως τα πράγματα, να αποκλείουν ορισμένους τομείς ή να προβλέπουν αιτιολογήσεις για ε, δημόσια πολιτική. Άλλο θα είναι μια καλή ιδέα να χαρακτηριστεί, να προβλεφθεί συγκεκριμένα η πρόσβαση στη διαδικασία. Για παράδειγμα, όπως είπα πριν, να εξαντλούνται τα εθνικές διαδικασίες πριν να μπορεί να προσφύγει ο επενδυτής στην ε, ε, διεθνή διατησία. Να αποκλείονται οι αβάσιμες προσφυγές και ούτω καθεξής, να υπάρχει διαφάνεια, κώδικας δεοντολογίας και μηχανισμός εφέσεων. Ε, εν συμπεράσματι νομίζω ότι από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι να παρέχεται πλήρης και ορθές, παρέχονται πλήρης και ορθές, και πληροφορίες. Νομίζω ότι οι νομοθέτες και αυτοί που ασκούν πολιτική και το κοινό έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν όλες τις πτυχές του συστήματος και μετά αποφασίζουν αν θα το συμπεριλάβουν ή όχι. Το να περιληφθεί κεφάλαιο για την προσθέτει των επενδύσεων στην TTIP έχει πολλά πλεονεκτήματα. Η ρύθμιση που προβλέπετε δεν είναι απαραίτητα τέλεια, αλλά γιατί να το πετάξετε όλο μαζί στα σκουπίδια. Μπορεί να βελτιωθεί. Μία συνολικά ρυθμισμένη ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η TTIP μπορεί να αποτελέσει και το μοντέλο και για μελλοντικέ συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με άλλες χώρες Εάν δεν περιληφθεί σύστημα αεστίας στη συμφωνία με τις ΗΠΑ, πώς θα πάει μετά στην Κίνα να πει ότι θέλει να βάλει εκεί σύστημα αεστίας. Μπορεί να δοθεί και ένα σημαντικό παράδειγμα που θα λειτουργήσει και ως καταλήτης για να βελτιωθεί η παγκόσμια ε, νομοθεσία προστασία των επενδύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ξεκάθαρο το μήνυμά σας. Απαιτείται βελτίωση. Ο τρίτος πανελίστ είναι ο κύριος James Ζαν, διευθυντής της Διεύθυνσης Επενδύσεων στην UNCTAD. Θα εστιάσει σε θέματα που σχετίζονται με τις επενδύσεις, τις επιχειρήσεις και την βιώσιμη ανάπτυξη. Προετοιμάζεται δε μία ετήσια έκθεση σχετικά. Κύριε Ζάν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μεγάλη μου τιμή που είμαι σήμερα προσκεκλημένο στο Ευρωκοινοβούλιο ώστε να κάνω μια παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Φαντάζομαι ότι το θέμα αυτό έχει συζητηθεί εκτεταμένα σε αυτό το πλαίσιο, οπότε εγώ θα ήθελα απλά να θυμίσω ότι το ISDS είναι ένας μηχανισμός επιβολής ένα εργαλείο ώστε να εφαρμόζονται οι ουσιαστικές διατάξεις διεθνών επενδυτικών συμφωνιών. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει κανείς να εξετάσει το ISDS απομονωμένα, αλλά σε σχέση με τις ε, ε, ουσιαστικές διατάξεις και τους κανόνες που προβλέπονται από τις διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες. Και υπάρχει σχέση ανάμεσα στις διατάξεις και τη διαδικασία και αυτή η σχέση θα πρέπει πάντοτε να είναι υπόψη μας όταν συζητάμε για μεταρρύθμιση του ISDS χωρίς ένα συνολικό πακέτο το οποίο θα ασχολείται τόσο με την ουσία των διεθνών επενδυτικών συμφωνιών όσο και με το ICS, οποιαδήποτε απόπειρα μεταρρύθμισης θα είναι κατακαιρματισμένη. Γι' αυτό και έχω προετοιμάσει μια γραπτή εισήγηση και θα ήθελα απλά να τονίσω κάποια σημεία κλειδιά, ειδικά αυτά που προσδιορίζεται στην ανακοίνωσή σας ενώ στη γραπτή μου εισήγηση εστιάζω σε τέσσερις πτυχές. Η μία είναι ο εντοπισμός των βασικών προκλήσεων που, έχουν να αντιμετωπίσουν, που έχει να αντιμετωπίσει το καθεστώς διεθνών επενδύσεων. Έπειτα να δώσω κάποια στοιχεία κλειδιά όσον αφορά την τρέχουσα χρήση του ISDS και τέλος να συνεχίσω τη σημερινή συζήτηση στα υπέρ και στα κατά των μηχανισμών ISDS ε, και τέλος, που είναι αυτό που είναι και το πιο σημαντικό μου τμήμα παρουσίασης, είναι να αναλύσουμε τις πιθανές επιλογές μεταρρύθμισης του ISDS καθώς και τις επιπτώσεις αυτών των επιλογών. Να πω εξ αρχής ότι το διεθνές ε, καθεστώς επενδυτικών συμφωνιών είναι εξαιρετικά περίπλοκο, αποτελείται από περίπου 3.000 3.260 επενδυτικές συμφωνίες σε διμερές, περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο. Ε, μέχρι τα τέλη δηλαδή του 2014, σύμφωνα με τις στατιστικές που έχουμε στη διάθεσή μας. Εντός αυτού του καθεστώτος, η ρύθμιση διαφορών είναι το πιο περίπλοκο στοιχείο και δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις ε, για γρήγορη ε, λύση. Για το Διεθνέ Καθεστώ επενδυτικών συμφωνιών υπάρχουν ε, συγκεκριμένες προκλήσεις. Η μία αφορά το χώρο πολιτικής, δηλαδή το δικαίωμα νομοθεσίας ε, ε, των εθνικών κυβερνήσεων. Δεύτερον είναι η ενσωμάτωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μέσα στις συμφωνίες τι επενδυτικές. Μέχρι στιγμής πολύ λίγες συνθήκες έχουν ενσωματώσει στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, πιο πρόσφατες μόνο το έχουν κάνει αυτό. Και η ε, τρίτη ευρεία πρόκληση είναι η συστημική πρόκληση λόγω του συστημικού, συστημικά περίπλοκου χαρακτήρα αυτού του τεράστιου σώματος ε, διεθνούς ε, νομοθεσίας, διεθνούς δικαίου. Πριν στραφώ σε πιθανούς τρόπους για τη μεταρρύθμιση του ISDS, θα ήθελα να τονίσω κάποια στοιχεία που είναι ουσιαστικά. Το σύνολο των γνωστών υποθέσεων ε, ρύθμισης διαφορών με βάση συμφωνίες ή συνθήκες ε, έχει φτάσει στις 608 μέχρι τα τέλη του 2014. Βλέπουμε λοιπόν μια αύξηση των υποθέσεων ετησίως. Όσον αφορά τα χώρες υποδοχής, οι περισσότερες ε, ε, καταγγελίες SDS ε, προέρχονται από επενδυτές από διάφορες χώρες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά το 50% όλων των υποθέσεων, ενώ αυτές που προέρχονται από τις ΗΠΑ ανέρχονται στο 22% των υποθέσεων. Όσον αφορά τις χώρες απάντηση, έχουμε 100 κυβερνήσεις που έχουν απαντήσει σε διαμεσολαβήσεις ιδιαιτησίες. 70% των γνωστών υποθέσεων έχουν ε, προέρθει, μάλλον ε, ε, καταγγελίες έχουν γίνει έναντι αναπτυσσόμενων οικονομιών ή οικονομιών που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. Αν το δούμε όλα αυτά από ευρύτερη προοπτική, έχουμε περίπου 26 3 εκατομμύρια δολάρια όσον αφορά την το, σε τι ανέρχονται τα στόκ αυτών των πολυεθνικών εταιριών και πρόκειται για 892.000 ε, θηγατρικές εταιρείες παγκοσμίω. Τεράστια τα νούμερα λοιπόν. Αν συγκρίνει κανείς ε, τις 608 μόνο υποθέσεις ε, διαθέτησης διαφορών δεν είναι και πολύ μεγάλος αριθμός. Στις δύο τελευταίες δεκαετίες κατατέθηκαν μονάχα 608 ε, τέτοιες ε, καταγγελίες. Ακόμα και αν έχουμε κάποιες άγνωστες υποθέσεις που υποθέτουμε ότι ανέρχονται στο ίμιση των γνωστών υποθέσεων, θα φτάναμε τις 800, πράγμα το οποίο είναι πάλι περιορισμένο νούμερο. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις πρόκειται για τομείς πολιτικής που είναι πολύ σημαντικοί και έχουν αντίκτυπο και όλα σε αυτούς τους τομείς, όπως ας πούμε ενεργειακή πολιτική, η πολιτική υγείας, ε, ε, δημοσιονομική κρίση και σε κάποιες περιπτώσεις πρόκειται και για τεράστια ποσά. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να αξιολογήσουμε πολύ προσεκτικά το κόστος και τα ωφέλη του ISDS και να σχεδιάσουμε ένα σύστημα για να τη ρύθμιση των ε, ε, διαφορών που αφορούν επενδύσει, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκε των επενδυτών, των κυβερνήσεων αλλά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Έχω και μια ανάλυση για τα υπέρ και τα κατά του ISDS. Ε, είναι γνωστή ανάλυση αυτή νομίζω και δεν χρειάζεται να την αναλύσω τώρα εδώ. Γι' αυτό και θα περάσω στο επόμενο κομμάτι της ε, παρουσίασής μου, δηλαδή ποια κατεύθυνση θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Η σημερινή συζήτηση για τα θέματα ESDS έχει ξεπεράσει το θέμα του, της ύπαρξης ή μη του συστήματος ESDS. Το θέμα είναι πώς θα προχωρήσουμε σε περίπτωση που αποφασίσουμε να εγκαταλείψουμε το ISDS και τι βελτιώσεις θα πρέπει να γίνουν στο ISDS έτσι ώστε, ε, μάλλον σε περίπτωση που αποφασίσουμε να το διατηρήσουμε το σύστημα αυτό. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με τη ρύθμιση των διαφορών εάν δεν υπάρχει το ISDS. Να ξεκινήσω λοιπόν με τις πιο άμεσες επιλογές. Δηλαδή, εάν, αν καταργηθεί τελείως το ESTS, τι παραμένει. Παραμένει η πρόσβαση των επενδυτών στις χώρες δικαιοδοσίες, στις χώρες υποδοχής, καθώς και στα όργανα ε, επίλυσης διαφορών που έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στα κράτη διμερώς. Αυτές θα είναι οι δύο επιλογές εάν δεν υπάρχει το σύστημα ρύθμισης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών. Τώρα, όσον αφορά την ε, εθνική δικαιοδοσία και την επίλυση διαφορών με βάση αυτήν, ήδη ε, ο πρώτος ομιλητής ανέλησε τα υπέρ και τα κατά, δηλαδή τις αδυναμίες του να βασίζεται κανείς μόνο στην εθνική ρύθμιση διαφορών. Δεν χρειάζεται λοιπόν να τα επαναλάβω εγώ αυτά τα υπέρ και τα κατά. Να πω μόνο ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα που εμπλέκονται εδώ. Το ένα έχει να κάνει με το επίπεδο του TTIP, δηλαδή σε ποιο βαθμό στην Ένωση το μόνιμο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα ήθελε να αναλάβει αυτή τη συνθήκη ή το ISDS ε εν γέννη. Αυτό είναι το ένα σκέλος της ερώτησης. Το άλλο είναι ότι για όλες τις ε, ενωτικές συνθήκες, δηλαδή η Ένωση δεν υπογράφει μόνο συνθήκες με τις ΗΠΑ, αλλά και με άλλες χώρες Ποιο θα είναι ο τρόπος για να αντιμετωπιστούν όλες αυτές όλο αυτό το περίπλοκο σώμα συνθήκων, επενδυτικών συνθήκων μέσω των εθνικών μηχανισμών ρύθμισης διαφορών. Υπάρχει δηλαδή κάποιος ε, περιορισμός όλα αυτά. Έπειτα έχουμε το δεύτερο σκέλος που είναι κράτος προς κράτος και ρύθμιση διαφορών. Είναι ο κλασικός τρόπος ε, ρύθμισης διαφορών σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Εκεί περιλαμβάνονται όλες οι διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες όπου περιλαμβάνεται αυτός ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών κράτους προς κράτος και εκεί περιλαμβάνεται και η προσέγγιση του ΠΟΕ. Δηλαδή ε, η ρύθμιση διαφορών ε, στις διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες. Γιατί λοιπόν να μην βασιστούμε αποκλειστικά σε αυτό το υπάρχον σύστημα, το ισχύον σύστημα. Το μόνο πλεονέκτημα είναι ότι θα μειώνονταν η έκθεση της χώρας υποδοχής στη διεθνή διατησία και ότι ένας επενδυτής θα είχε φυσικό συμφέρον να διεκδικήσει τα δικαιώματά του στην χώρα του στη χώρα προέλευσής του. Και θα έπρεπε να σκεφτεί κανείς και τις ευρύτερες πολιτικές επιπτώσεις του να κατηγορήσει κανείς μια χώρα ότι παρεβίασε τη διεθνή νομοθεσία. Πρόκειται για μια μεγάλη αδυναμία δηλαδή της διετησίας χώρας προς χώρα και οι επενδυτές θα εξαρτώνταν απόλυτα από την επιθυμία και την καλή θέληση της χώρας υποδοχής να παρέμβει. Και βέβαια για τους μικρομεσαίους επενδυτές θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Θα έπρεπε δηλαδή να πείσουν τη χώρα υποδοχής ότι η παραβίαση της λόγω συνθήκης επενδυτικής συμφωνίας είναι τόσο σημαντική που θα επηρεάσει τις εξωτερικές της σχέσεις. Σε πολλές περιπτώσεις θα ήταν άδικο, άδικη μάχη, χαμένη μάχη, ειδικά για τους μικροεπενδυτές. Έπειτα, χώρα προς χώρα και σχετική ε, διατησία. Σε περίπτωση εμπορίου, μία διαφορά ήδη έχει επιπτώσεις για την οικονομία μιας ολόκληρης χώρας, ενώ όταν πρόκειται για μία επενδυτική διαφορά, συνήθως πρόκειται για ένα συγκεκριμένο μόνο επενδυτή. Άρα, η χώρα, το κράτος, είναι πιο λίγο απίθανο να διεκδικήσει κάποια διετησία σε ένα εμπορικό θέμα αντί σε ένα επενδυτικό θέμα. Τελειώνοντας, δεν νομίζω ότι η πλήρης κατάργηση του ESDS ε ή η απόλυτη εξάρτηση από ε, μηχανισμούς επίλυσης διαφορών εκτός του ESDS ε μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Πρέπει ωστόσο να αντιμετωπίσουμε τις θεμητές ανησυχίες όσον αφορά την λειτουργία του ESDS, εάν ληφθεί απόφαση να διατηρηθεί το σύστημα αυτό. Και έτσι έρχομαι στο δεύτερο τμήμα της παρουσίασής μου σε σχέση με τις επιλογές για μεταρρύθμιση του ISDS. Η Άγκτα έχει μελετήσει το θέμα εδώ και χρόνια και επίσης έχει συνοψίσει την συζήτηση που γίνεται παγκοσμίω και έχουμε καταλήξει σε πέντε επιλογές μεταρρύθμισης. The, the, five, uh, the five reforms options include limiting investors' access to ISDS and improving procedures in existing international convention, uh, conventions dealing with ISDS, such as the Convention on the Center of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 investment regime to ensure the consistency. And overall, we need a new generation of IAs that address the challenges of investment policies of the 21st century. Thank you very much. Thanks a lot. And now, last but not... Ευχαριστώ και τελευταίος αλλά όχι ίστατος, ο καθηγητής Στέφεν Χίντεν Λάγκ από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Θα μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση για μια μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Expo που έλαβε χώρα το 2014 με τον καθηγητή Κιούπερ, τον κύριο Γιάνσεν και τον ίδιο τον κύριο Χίντεν Λάγκερ. Έχετε το λόγο λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να παρουσιάσω εν συντομία τα κύρια απορίσματα των τριών αυτών μελετών για την ε, διαθέτηση διαφορών επενδυτών κρατών που έγινε μετά από αίτηση της Επιτροπής ΙΝΤΑ πέρσι. Οι τρεις μελέτες έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν να υπάρξει μια αντικειμενική αντιμετώπιση της τωρινής συζήτησης για την επενδυτική προστασία στη Συμφωνία ΣΥΤΑ, Συμφωνία με τη Σιγκαπούρη και την ΤΙΤΙΚ. Να ξεκινήσω αμέσως με αυτά τα οποία θεωρώ ότι είναι τα πιο σημαντικά μηνύματα των τριών μελετών που τα σημερινές τρεις μελέτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει σύγχρονα κεφάλαια επενδύσεων σε όλες τις ε, πλήρες τις συνολικές συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου ή όταν αυτό είναι απαραίτητο θα πρέπει να διαπραγματευτεί χωριστές συμφωνίες επενδυτικού χαρακτήρα. Οι ουσιαστικές δεσμεύσεις θα πρέπει να υποστηρίζονται από ένα μηχανισμό επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών. Με το να γίνει κάτι τέτοιο με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έκανε μια σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου στον τομέα αυτό και συγχρόνως θα προστάτευε τις ευρωπαϊκές επενδύσεις. Στο βαθμό που οι μελέτες έχουν ήδη εξετάσει την ε, Συμφωνία ΣΥΤΕ, ε, ε, θεωρούν ότι έχει υπάρξει μεγάλη πρόταση, πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσουν αυτό το καθεστώς. η ΣΥΤΑ είναι μια καινο, καινοτόμος συμφωνία γιατί δημιουργεί μια νέα ποιότητα στην αντιμετώπιση τέτοιων διαμαχών. Ξεκινάει από αμερικανικά και καναδικά μοντέλα και αναπτύσσει αυτά τα πρότυπα με πιο πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Υπάρχει το <clears throat> δικαίωμα για τη ρύθμιση και γίνεται σαφέστερη η διαδυσία μεταξύ κρατών και ε, επενδυτών και επομένως λιγότερο μεροληπτική. Παρά το γεγονό λοιπόν ότι αναγνωρίζουμε την πρόοδο η οποία επιτεύχθη με τη ρυθμιστική προσέγγιση τη ΕΤΑ, έχουμε πέντε σημαντικέ προκλήσει που παραμένουν. Τέσσερι από τι πέντε είναι περιοχές που έχουν αναφερθεί και από τον κύριο Μπέρκ στην ε, έκθεση της Κομισιόν για τη δημόσια διαβούλευση σε σχέση με το ISDS στη Συμφωνία CHI-CHIP. και οι ουσιαστικές αυτές ε, ρήτρες δεν περιλαμβανόντουσαν στο περιεχόμενο της μεθελέτης μα. Πρόκειται για τι εξής προκλήσεις. Η, το κείμενο της ΣΥΤΑ δεν συμπεριλαμβάνει παρά μόνο ανεπαρκώς τα εθνικά νομικά συστήματα και αποδυναμώνει λειτουργικά συστήματα όπως είναι το Ολλανδικό ή το Γαλλικό παραδείγματος χάρη. Η ενίσχυση του διεθνού δικαίου στο διεθνή τομέα σε κάποιο βαθμό σημαίνει παράλληλα αποδυνάμωση του εθνικού δικαίου. Δεύτερον, το κείμενο της ΣΥΤΑ δεν δημιουργεί ένα εφετείο, αλλά απλώς ασαφώς αναφέρεται σε κάτι τέτοιο. Τα νομικά σφάλματα ή τα σφάλματα ουσίας ή οι συγκρουόμενες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια της ΣΥΤΑ δεν μπορούν να τύχουν αποτελεσματικής θεραπεία. Η συνεκτικότητα στην ερμηνεία και την εφαρμογή αυτής της συνθήκης λοιπόν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί. Τρίτον, το κείμενο της ΣΥΤΑ δεν διασκεδάζει την ε, εντύπωση του κοινού ότι τα δικαστήρια θα είναι μεροληπτικά υπέρ των επενδυτών. Οι διαδικασίες θα ξεκινούν σχεδόν πάντα από τους επενδυτές και οι διαιτητές μπορούν να αλλάζουν συνέχεια τους κανόνες και μπορεί κανείς να τους κατηγορήσει ότι έχουν σύγχρονους συμφερόντων, ότι έχουν μια φιλική προς τους επενδυτές ε, λήψη απόφασης. Τέταρτον, το κείμενο της ΣΥΤΑ αφήνει τα διοικητικά θέματα, τα οποία μπορεί να είναι πολύ σημαντικά για τις ε, διαδικαστικές αποφάσεις, όπως παραγωγός χάρη η επιλογή των διαιτητών, τα αφήνει σε μια γραμματεία ενός ε, φορέα, διεθνούς φορέα, όπου οι ευρωπαϊκές αρχές δεν έχουν μεγάλη επιρροή. Και τελευταίο, αλλά όχι το ίστατο, ο μηχανισμός που περιλαμβάνεται στην Συμφωνία ΣΥΤΑ για την επίλυση διαφορών ενδέχεται να μην είναι συμβατός με τις ευρωπαϊκές συνθήκες, γιατί δεν περιλαμβάνει τη δυνατότητα πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και δεν σέβεται την αρχή της αυτονομίας του Ευρωπαϊκού Δικαίου αυτό το οποίο χρειάζεται αντίθετα. Η Ευρώπη είναι ένα ανεξάρτητο και καινοτόμο υπόδειγμα ESDS που να προστατεύει τους επενδυτές και να σέβεται τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της. Ένα ευρωπαϊκό μοντέλο μπορεί να προστατεύσει τις ε, επενδύσεις στο εξωτερικό με ένα υφόρο τρόπο και έτσι να θεσπίσει ε, παγκόσμια πρότυπα για τις επενδύσεις θα έφερνε με τον τρόπο αυτό σε μια σχετική ισορροπία τα συμφέροντα των επενδυτών και των κρατών μελών, αλλά συγχρόνως με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διατηρώντας την νομική παράδοση και τις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα τέτοιο ευρωπαϊκό μοντέλο θα έπρεπε να ενσωματώνει επαρκώς την ε, λειτουργία των εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων στην επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών μελών γιατί τα εθνικά αυτά συστήματα έχουν τα βασικά, βασικά δικαιώματα και τα εφαρμόσουν αποτελεσματικά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το να, έχουν ελαστική, να υπάρχουν ελαστικοί κανόνες τοπικής θεραπείας, τοπικής απόφασης, που να εξαρτώνται από τις αρμοδιότητες των εθνικών συστημάτων δικαιοδοσίας σε διάφορες περιπτώσεις. Η υποχρέωση της εξάλλησης των τοπικών ε, βαθμών δικαιοσύνης μπορεί να βασίζεται σε ένα εύκαμπτο σύστημα που έχει να κάνει με τι αρμοδιότητε δικαστήριων. Δεύτερον, ένα τέτοιο ευρωπαϊκό υπόδειγμα θα πρέπει να δημιουργήσει ένα μόνιμο εφετείο για διαφωνίε αυτού του είδου όταν δεν μπορούν να επιληθούν επί τη βάση διαιτησίας για μια συμφωνία αλλά επίσης θα μπορεί να είναι ανοιχτό και για διατησία σε περίπτωση συμφωνιών προς τρίτες χώρες. Τρίτον, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο μπορεί να μειώσει, να καταπραίνει την, τον φόβο ότι υπάρχει μεροληπτικός χαρακτήρας υπέρ των επενδυτών στα διαιτητικά δικαστήρια. Αυτό να μπορεί να γίνει με αύξηση των δυνητικών διαιτητών οι οποίοι μπορούν να διοριστούν για μια διαδικασία διαιτησίας επί τη βάση της εγγραφής του σε ένα κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να είναι ανοιχτός σε όλους τους ε, δικηγόρους οι οποίοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα για διαιτησία αυτού του είδους. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να πάψει να υπάρχει διαιτησία ad hoc και να υπάρχει άσκηση κρατικής εξουσίας από ένα μόνιμο δικαστήριο. Τέταρτον, το ευρωπαϊκό μοντέλο θα πρέπει να κάνει εξουσιοδότηση για διοικητικές ε, αποφάσεις σε διεθνείς φορείς οι οποίοι να έχουν έδρα στην Ευρώπη ώστε να δίνουν μια ουσιαστική εξασφάλιση της ε, σωστής τους λειτουργίας ως διεθνών φορέων. Αν εναλλακτικά δεν πρέπει να υπάρχει καμία απόλυτα διακριτική ευχέρεια του επικεφαλής του φορέα διαιτησίας σε σχέση με τη ΣΥΤΑ ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία. Πέμπτον, ένα ευρωπαϊκό υπόδειγμα θα πρέπει να εξασφαλίζει σε επαρκή βαθμό την αυτονομία του ευρωπαϊκού δικαίου και το μονοπόλιο σε δικαστικά θέματα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν προστατευτεί το ευρωπαϊκό δίκαιο από την δυνατότητα επιμόλυνσής του από διαδικασίες διευθυνσίες. Όταν προκύπτουν θέματα ευρωπαϊκού δικαίου σε μια διαδικασία διαιτησίας, θα πρέπει ενδεχομένω να εμπλέκεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να υπάρξουν δεσμευτικέ ερμηνείε. Για να μην υπάρχουν αμφισημίε, θα πρέπει ένα κείμενο ISDS σε μια συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για γνωμοδότηση νομικά, σε νομικό επίπεδο προτού συμφωνηθεί ή έστω και εφαρμοστεί. Γενικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταφέρει να ε, ενημερώσει τη Συμφωνία ΣΥΤΑ και να τη φέρει σε επίπεδο του, της, των ρυθμίσεων της Βόρειας Αμερικής και έχει βελτιώσει τη συμφωνία των κρατών μελών. Αλλά υπάρχουν χώροι για περαιτέρω βελτίωση. Εφόσον δεν έχει συναυθεί ακόμα μια συμφωνία για τα θέματα αυτά, υπάρχει μια ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό και βιώσιμο μοντέλο για επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών μελών που θα λειτουργήσει σαν υπόδειγμα για τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πάρα πολύ ε, επακριβή αυτά που είπατε. Έχουμε τώρα την διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων από τα μέλη μας, περίπου 20 λεπτά. Σας παρακαλώ να είστε σύντομοι και περιεκτικοί. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε ερωτήσεις και όχι δηλώσεις. Ερωτήματα λοιπόν παρακαλώ και να εξηγείτε σε ποιον απευθύνεται το ερώτημα το οποίο θέλετε να θέσετε. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για τη διαδικασία μας. Έχουμε ένα ανοιχτό κατάλογο. Ξεκινώ με την Έμα Μακλάρεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους αυτούς οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στο πάνελ μας σήμερα το απόγευμα. Το μυαλό μου αρχίζει να υπερθερμαίνεται άμα σκεφτούμε όλες αυτές τις δυνατότητες που υπάρχουν και που ανοίγονται ενώπιόν μας. Αυτό το οποίο είναι σαφές και έχει γίνει σαφές σήμερα το απόγευμα είναι ότι είναι απαραίτητη η προστασία των επενδυτών με κάποια μορφή. Δεν είναι απλή λύση να πούμε ότι δεν θα έχουμε προστασία των επενδυτών. Αυτό είναι απαραίτητο και μπορούμε να δούμε από τι στατιστικέ που μα παρουσιάσαν σήμερα το απόγευμα ότι είναι οι επενδυτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση που χρειάζονται αυτή την προστασία περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Θα πρέπει να δούμε τώρα πώ μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση και να λάβουμε υπόψη τι προτάσει που ακούσαμε σήμερα το απόγευμα για να βελτιώσουμε την υπάρχουσα μορφή του ISDS που έχουμε σήμερα ώστε να υπάρχει η προστασία αυτή και να είναι βελτιωμένη προστασία. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να αντιμετωπίσουμε την περιορισμένη πρόσβαση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα δικαστήρια. Μερικές από τις λύσεις που προτείνω θα κάνουν ακόμα πιο μακροχρόνια, ε, πολυδάπανη και πολύπλοκη τη διαδικασία αυτή. Εμείς αντίθετα θέλουμε να βοηθήσουμε αυτούς οι οποίοι χρήζουν προστασίας να νιώσουν ότι μπορούν να επενδύσουν. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνήσουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή τη ε, διαδικασία με το να υπάρχει δυνατότητα έφεσης, να βελτιώσουμε σε σχέση με τη ΣΥΤΑ το κείμενο για την ε, προστασία των επενδυτών. Και θέλω να θέσω ένα ερώτημα στον τελευταίο μιλητή, ο οποίος μας έδωσε την εντύπωση ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερο για το ISDS για να διασκεδάσουμε την άποψη του κοινού ότι μια τέτοια διαδικασία θα αποβεί υπέρ των επενδυτών. Είναι απαραίτητο να αποφύγουμε τη δημιουργία μιας τέτοιας εντύπωση στην κοινή γνώμη, αλλά ίσω θα έπρεπε να μα εξηγήσει ο κύριο καθηγητή καλύτερα με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, πέραν της, ε, του να βασίζονται όλα αυτά στο δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα Σας ευχαριστώ. Εγώ βεβαίω ε, θα παίξω σύμφωνα με τον κανόνα, δηλαδή δεν θα κάνω δήλωση, αλλά ερώτηση θα υποβάλω. Πρώτη προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριο Μπράουν. Όταν λέτε ότι στη δημόσια διαβούλευση υπάρχουν μάλλον επιφυλακτικές απαντήσεις, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι το 97% των απαντήσεων, όχι 51% ούτε 62%, 97% των απαντήσεων είναι αρνητικές απέναντι στο σύστημα EDS. 150.000 πρόκειται για 145.000. Ερώτηση, διότι ένα από τα διακυβεύματα βεβαίως και όλοι συμφωνούν για την προστασία των επενδύσεων και ότι η προστασία των επενδύσεων σε κάποια φάση μπορεί να οδηγήσει στην αμφισβήτηση μιας απόφασης των κρατών ή των περιφερειών ή των ε, νόσων ή του ομοσπονδιακού επίπεδου. Όμως θα πρέπει να διαρωτηθούμε ποιος είναι σε θέση να ε, διαιτητεύσει. Είναι οι, δικαστε... Ε, είναι οι δικηγόροι, τα ιδιωτικά δικαστήρια κριτήρια είναι οι εθνικές δικαιοδοσίες. Άρα τίθεται το ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων. Για παράδειγμα, η κυρία Μπαϊτάς, η οποία παρενέβη ως καθηγήτρια δικαίου που έχει συμβουλεύσει κυβερνήσεις, μπορεί να μας επιβεβαιώσει ότι εργάζεται επίσης και για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Χημικής Βιομηχανίας και για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν εξαρτήσεις υπέρ του ISDS. Επόμενος ε, μιλητή ήταν ο εκπρόσωπος της ΑΝΚΤΑΝΤ, ε, η Κνούσεντε στα γαλλικά. Στις 4.000 επενδυτικές συμφωνίες ή πάση περιπτώσει όσες υπάρχουν, πόσες εκπνέουν αυτή τη στιγμή. Γιατί πιστεύω ότι εφόσον θέλουμε να αναπτύξουμε μια στρατηγική επενδυτική, θα πρέπει να γνωρίζουμε επίσης ποιο είναι ο χώρος μας για να το κάνουμε αυτό. Και έπειτα στον τελευταίο μιλητή θα ήθελα να πω ότι είπε πως τουλάχιστον τρεις χώρες με το ISDS βλέπουν να έχει αποδυναμωθεί το δικαστικό του σύστημα. Ε, κάτω νομίζω είπε Γαλλία και άλλη μια χώρα, ε, μπορεί να μας πει αν τελικά υποστηρίζουν το ISDS ή όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σούστερ. Έχω τρεις ερωτήσεις. Αφενός ελέγχει ότι το ISDS υποτίθεται θα προωθήσει κιόλας τις επενδύσεις θα κινητοποιήσει. Υπάρχει καμιά στατιστική των τελευταίων 10-15 ετών σχετικά με επενδύσεις που δεν έγιναν μεταξύ Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου δεν υπάρχει ISDS, διμερείς ISDS. Υπάρχουν στατιστικές, λοιπόν, και σχετικά με άλλους λόγους που οδήγησαν ώστε να μην γίνουν κάποιες επενδύσεις. Απευθύνομαι ιδίως στην κυρία Μπάτενς και στον ε, εκπρόσωπο της Κομισιόν άκουσα και ορισμένα αντιφατικά πράγματα. Αφενό να εξαντληθεί, λέει, να εξαντληθούν μάλλον οι εθνικοί βαθμοί δικαιοδοσία. Ταυτόχρονα η κυρία Μπέρτεν, αλλά αν κατάλαβα καλά και ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπαν ότι τα εθνικά δικαστήρια εν μέρη δεν μπορούν καν να είναι αρμόδια. Αν όμως δεν είναι αρμόδια τα εθνικά δικαστήρια, δεν είναι τότε νοητό να μπει μέσα στην TTIP, να συμφωνηθεί δηλαδή μέσα στην TTIP ότι οι χώρες μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν, θα πρέπει να προβλέψουν νομοθετικές ρυθμίσεις που θα εξισώνουν τον αλλοδαπό επενδυτή με τον ημεδαπό. Και τελευταία ερώτηση για τα διεθνή εμπορικά δικαστήρια. Θέμα όπου δεν συμμετέχουν ανεξάρτητοι δικαστές και ότι αυτοί οι δικαστές θα πρέπει να πληρώνονται αναϋπόθεση. Το επιχείρημα είναι τώρα ότι τα δικαστήρια αυτά είναι τόσο δαπανηρά. Ε, μα υπάρχει κανένα, καμία στατιστική που, ε, που δείχνουν πόσο δαπανηρότερα είναι αυτά τα δικαστήρια σε σχέση με ιδιωτική διατησία Χάιντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και ιδέες σχετικά με το πώς μια βελτιωμένη εκδοχή της ISTS θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Να επανέλθω σε αυτά που ο κύριος Ζάνη και να του θέσω μια ερώτηση. Έκανε μια σημαντική παρατήρηση. Είπε δηλαδή ότι ο μηχανισμός ε, ρύθμισης ε, διαφορών δεν θα πρέπει να είναι ξεχωριστός από τα υπόλοιπα τμήματα. Αυτό εδώ μου φαίνεται ότι αν μιλούμε για την TTIP, όπου απέχουν πολλοί αμερικανικές από τις ευρωπαϊκές θέσεις, για παράδειγμα σχετικά με το policy space, όπως το είπαν και πολλοί από τους ομιλητές, θα ήθελα ο κύριος Ζαν και η Δόκτωρ Μπάτινς να μου απαντήσουν στο εξής. Εάν βασιζόμαστε στον ΠΟΕ και στο άρθρο 20 του ΚΑΤ για τις γενικές εξαιρέσεις που αναφέρονται στον χώρο πολιτικής, στο της πές. οι χώρες μέλη δεν θα αντιμετωπίζουν την πρόκληση να αιτιολογούν τα μέτρα πολιτικής που λαμβάνουν απέναντι στην προστασία του επενδυτή και ποιες είναι οι εμπειρίες από τα πάνελ του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Δεύτερο, ο καθηγητής Χίντελανγκ είπε ότι η ISDS ίσως να μην είναι απόλυτα συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ορισμένοι παρακολουθήσαμε την πρόσφατη απόφαση της 8 Δεκεμβρίου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την μη συμβατότητα της πρόσβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Υπάρχουν κάποιες νομικές αρχές που, μπορούν, ε, που μπορεί να απορρέουν από την απόφαση αυτή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και μήπως το ίδιο αναλογικά μπορεί να εφαρμοστεί και στην περίπτωση της αγιστίας. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Έχω ακόμα 7 εγγεγραμμένους. Σήκω. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι σε σχέση με τη... τα όσα μας παρουσίασαν οι σημερινοί μιλητές, θα ήταν σημαντικό να κατανοήσουμε καλύτερα εάν έχουμε φτάσει στη διατύπωση μιας βελτιωτικής πρότασης ε, όσον αφορά τον θεσμό αυτό, διότι σε σχέση με τις ενδείξεις περιορισμένων υποθέσεων επί των οποίων εφαρμόζεται, σε σχέση με τις απαντήσεις που τείνουν να ε, οδηγούν προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή είδαμε ότι δεν θέλουμε να παρέμβουμε ή να υποκαταστήσουμε τα δικαστήρια ή τα, εθνική, την εθνική νομοθεσία. Θέλουμε να προσφέρουμε ε, ε, βεβαιότητα δικαίου ιδιαίτερα όσον αφορά την κατάσχεση του, της ιδιοκτησίας ή την μειονεκτική ενδεχόμενα θέση που μπορεί να βρεθεί ένας ξένος επενδυτής σε σχέση με κρατικές εταιρείε. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι πρέπει να κατανοήσουμε ποια θα ήταν η διατύπωση μιας βελτιωτικής πρότασης, δηλαδή με έναν κώδικα συμπεριφοράς, με ε, Καταλόγου συγκεκριμένους ε, για τις διάφορες βαθμίδες ε, δικαιοδοσίας. Εγώ είμαι κατά της ύπαρξης έφεσης. Η βεβαίωση βελτιωτικής πρότασης είναι από τη στιγμή που μια συμφωνία δίνει σαφήνεια σε μια απόφαση η οποία είναι τελεσίδικη γιατί διαφορετικά διατρέχουμε το κίνδυνο να χρησιμοποιήσουμε εκείνους τους συνηθισμένους μηχανισμούς που είναι διαρκώς επαναληπτικοί και απλώς ε, μακραίνουν τη διαδικασία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέω κύριο Σάντερσον. Ένα σημαντικό στοιχείο της συζήτησης για το ISDS είναι ότι υποτίθεται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων. Από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχουν εμπειρικά στοιχεία που να κατεδεικνύουν ότι κάτι τέτοιο λαμβάνει η χώρα. Θα ήθελα να μάθω από τους εμπειρογνώμονες αν συμφωνούν με αυτή την ιδέα. Νομίζω ο κύριος Ζαν θα είναι ο καταλληλότερος για να απαντήσει αυτό το ερώτημα. Ευχαριστώ. Κύριος Κάστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρία ερωτήματα. Ακόμα και αν πιστεύει κανείς ότι είναι σωστό οι επενδυτές να προστατεύονται οι επενδυτέ των εταιριών να προστατεύονται, γιατί δεν υπάρχει καμία μνήμα να δυνατότητας προστασίας των εργαζομένων όταν θίγονται τα δικαιώματά τους ή όταν πρόκειται για παραβίαση των δικαιωμάτων των καταναλωτών ή παραβίαση των ε, κανόνων για το περιβάλλον. Δεύτερον, ο κύριος Μπρός από την ε, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τη Γερμανία, ένα δικαστή του Συνταγματικού Δικαστηρίου στο παρελθόν, είχε πει ότι οι ιδιωτικέ διαδικασίες διαιτητικού χαρακτήρα δεν συνάδουν ούτε με το Σύνταγμα της Γερμανίας, ούτε με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν παραβίαση του διεθνούς δικαίου μια τέτοια συμφωνία. Και επίσης το θέμα που ανέφερε προηγουμένως ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν. Είναι έγκυρε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αυτέ οι διαδικασίε. Και τρίτον, οι διαδικασίε προστασία των ε, ε, επενδυτών μήπως θα οδηγήσουν και σε πολιτική πίεση στις κυβερνήσεις να καταλήγουν σε ορισμένες συμφωνίες. Στην περίπτωση της ναύτα, δηλαδή αμερικανικές εταιρείες έχουν ε, ουσιαστικά ε, στραφεί κατά των καραδικών αρχών γιατί απαγόρευσαν την υδρορογμάτωση. Ευχαριστώ. Και εγώ θα είμαι σύντομος και πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει να απάντηση των ερωτήσεων. Τα πρώτα ερωτήματα είναι αν έχετε παραδείγματα περιπτώσεων όπου οι επενδυτές στις ΗΠΑ έχουν τύχει διακρίσεων λόγω έλλειψης ISDS ή μη συγχρόνου ISDS και αν έχετε κάποιες εναλλακτικέ δυνατότητες για να υπάρξει προστασία των επενδυτών μας στις ΗΠΑ, ιδίως μικρομεσαίων <clears throat> επιχειρήσεων. και επίσης αν έχουμε επιστημονικά στοιχεία. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, μόνο με παραδείγματα μπορεί να καταλήξει κανείς σε, κάποιες, ε, ε, σε κάποιες συμπεράσματα. Κύριε Τούντερ, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Τρία σύντομα ερωτήματα. Στην ανάλυση κόστος ωφέλους, που, στην οποία αναφέρθηκαν πολλοί ομιλητές, δεν υπήρχε πουθενά το κόστος της ε, ρύθμισης που το ξέρουμε τώρα στην περίπτωση χάρη των συσκευασιών, των απλών συσκευασιών σε ορισμένε χώρε. Πώ θα πρέπει λοιπόν να το λάβετε αυτό υπόψη, και υπάρχουν ορισμένε χώρε επίση, οι οποίε έχουν κινηθεί σε μια διαφορετική κατεύθυνση και αποφάσισαν να μην ακολουθήσουν ένα σύστημα τύπου ISDS ή έχουν κάνει συμφωνίε που δεν εμπεριέχουν το ISDS, η Αυστραλία, Ηνωμένε Πολιτείε. Υπήρξε κάποιο αντίκτυπο αρνητικό για τι ροέ επενδύσεων Υπάρχει κάποιος αντίκτυπος που μπορείτε να πείτε ότι ήταν σημαντικός <clears throat> και μείωσε τις ε, εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών και για την TTIP και το ISDS. Κανείς δεν το έχει αναφέρει, αλλά οι Ηνωμένε Πολιτείε έχει, έχει εφαρμόσει πολλές φορές διεθνείς συνθήκες με εσωτερική νομοθεσία, γιατί αυτό δεν μπορεί να ισχύσει και για την προστασία των επενδυτών για να εξασφαλιστούν ότι οι αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων θα είναι πιο αποτελεσματικέ. Ο Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, και εσάς κύριε Πρόεδρε και για τις εισαγωγικέ παρατηρήσεις των ε, διαφόρων εμπειρογνωμόνων. Με έχουν καλύψει ορισμένοι συνάδελφοι σε άλλε ερωτήσεις, γι' αυτό έχω ακόμη τρει προς τον κύριο Ζαν. Πού βλέπετε να εντοπίζεται η αιτία για την δραματική αύξηση διαιτητικών διαδικασιών τα τελευταία χρόνια. Με τι συνδέονται. Είτε πρόκειται για διμερείς, είτε πρόκειται για πολυμερείς συμφωνίες που θεσπίζουν διαιτητικές διαδικασίες. Για δραστηριότητες επενδυτών. Είναι ανεπαρκείς οι ρυθμίσεις αυτές. γιατί αυξάνονται οι διαιτητικές διαδικασίες. Δεύτερο ερώτημα. Προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Χίντελανγκ είπε ότι στην προστασία επενδυτών στη ΣΕΤΑ δεν περιλαμβάνεται επαρκώς οι εθνικές νομοθεσίες και ότι είναι ασαφώς ορισμένες. Όμως πρόκειται για συμφωνία η οποία έχει μονογραφηθεί. Πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτό. Τρίτη ερώτηση για τον κύριο Ζαν πάλι. Πώς φαντάζεστε την δόμηση αυτού του Διεθνούς Διευθυντικού Δικαστηρίου στη βάση για παράδειγμα των όσων προβλέπονται για την ΆΝΚΤΑΤ και άλλους οργανισμούς των ΗΠΑ. Πρόεδρος Λάγκε, θα πρέπει τώρα να κλείσουμε το πρώτο αυτό τμήμα γιατί είναι τέλος πάντων και θέμα ε, δικαιοσύνης. Ε, γι' αυτό, αλλά έχω δύο ακόμη, η κυρία Κέλλερ και τον κύριο Λιμπρέρι, αλλά πρώτα η κυρία Κέλλερ σύντομα. Κυρία Μπάτενς, είπατε ότι θα μας δώσετε μια πρακτική οπτική πρακτική. Πόσα κερδίζει ένας δικηγόρος σε αυτές τις διαιτητικές διαδικασίες. Και μια δικηγορική εταιρεία όπως η δική σας, κατά πόσο εξαρτάται από το εισόδημα από αυτές τις υποθέσεις. Τώρα, ερώτηση για άλλον ομιλητή, αλλά δεν είμαι βέβαια για ποιον. Πάντως διαρωτώ με, εάν δώσουμε στους επενδυτές το δικαίωμα να προσφεύγουν κατά των κυβερνήσεων επειδή υφίσταται διακριτική μεταχείριση. Τι γίνεται με τους πολλούς ανθρώπους που βλέπω στην Αλοδαπή να υφίσταται διακριτικές μεταχειρήσεις στα ανθρώπινα δικαιώματά τους και δεν μπορούν να προσφύγουν κατά των επενδυτών είναι όμως ευθύνη των κυβερνήσεων να τους προστατεύσουν. Μήπως έχετε κάποια ιδέα σχετικά. Εσείς κύριε Ζαν, Νομίζετε ότι μεταρρυθμίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επαρκής και είναι σωστό να πει κανείς ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις περισσότερες υποθέσεις αυτό είναι καλό ή μήπως παρεμποδίζει αναπτυσσόμενες χώρες από το δικαίωμά τους να αναπτυχθούν. Και πώς αυτές οι υποθέσεις της δεν είναι γνωστές. Είπατε, ότι, είπατε κύριε ότι η ε, συμφωνία ΣΕΤΑ παίζει πρωτοποριακό ρόλο, αλλά δεν είχε η προηγούμενη ISTS. Τέλος, ο κ. Δημητρών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ τους τέσσερις ομιλητές που ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντες. Το θέμα δεν είναι αν πρέπει να προστατευτούν οι επενδυτέ, αλλά πώ θα πρέπει να προστατευτούν. Τρει λύσει προτάθηκαν. Πρώτον, αυτή τη Κομισιόν, δηλαδή διευθυνσία μέσω των κρατών. Δεύτερον, διεθνή διατησία ανάμεσα σε κράτη. Και τρίτον, εθνική δικαιοσύνη. Κανεί δεν υπερασπίστηκε τη δεύτερη λύση, άρα λοιπόν θα την αγνοήσουμε σιωπηρά. Ενώ τρει ομιλητέ μίλησαν υπέρ τη λύση πρώτων η Κομισιόν. Ωστόσο, εμένα μου δημιουργεί δύο ερωτήματα. Πρώτον, προ τον κύριο Ζαν, είναι πραγματικά υπέρ αυτή τη λύσης ε, διατησία ανάμεσα σε επενδυτέ και κράτη, γιατί μου φάνηκε πω έδειξε κάποιους δισταγμούς ε, για την υπεράσπιση αυτή τη λύση στο τέλο τη παρέμβασή του. Και η δεύτερη ερώτηση προ τον καθηγητή Ιντελάγκα, Εκείνο αν κατάλαβα προτιμά το πρότυπο των εθνικών δικαιοδοσιών, θέλει επίση να διατηρηθεί η αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά σε κάποια φάση αφήνει κάποιο χώρο στη διατησία και ομολογώ ότι δεν κατάλαβα πολύ καλά πώς όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Άρα λοιπόν ερώτηση, ποιο χώρο δίνεται στην διαιτησία στο δικό σας σχήμα, το μοντέλο που προτείνετε. Μάλιστα, ευχαριστώ. Και τώρα τρία λεπτά κάθε ειδικό. Κύριος Σλίγγελ Μίρλικ. Θα κάνω ό,τι μπορώ, πάρα πολύ σύντομα, με την κυρία Μακλάρεν. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Με τις ε, μικρομεσαίες στον Καναδά, υπήρχε η δυνατότητα για μια απλούστερη διαδικασία διατησίας και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ξαναδούμε. Για τον κύριο Σαντό, για τη διαδικασία διαβούλευση στην αλήθεια, δεν το κρύβω ότι 145.000 από 150 είπαν δεν μας αρέσει η TTIP και ή δεν μας αρέσει η ISDS. Για το θέμα της αμεροληψίας, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν έχει τέτοιου κινδύνους και οι κανόνες τώρα που έχουμε τώρα περιλαμβάνουν την αποκάλυψη δραστηριοτήτων κτλ. ώστε να ξέρει κανείς από πού προέρχεται κανείς και η σκούφια του επίσης. <clears throat> το θέμα των εθνικών δικαστηρίων. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και φυσικά και η σχέση με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Να είμαστε σαφείς και πάλι. Ακόμα και οι ευρωπαϊκές αποφάσεις του δικαστηρίου λένε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις διεθνείς ε, υποχρεώσεις, το κάνουμε για ανθρώπινα δικαιώματα και για άλλες συμβάσεις όπως είναι ο ΠΟΕ. Εδώ το θέμα είναι ότι τα δικαστήρια του ISDS δεν κοιτάζουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοιτάζουν τις διεθνείς υποχρεώσεις. Και φυσικά θα πρέπει να αφασίσει και αυτό το κοινοβούλιο ποιες είναι οι διεθνείς υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνουν. Το θέμα τώρα των στατιστικών, του κόστους και αν παροτρύνει τις επενδύσεις. Φυσικά οι αποβάσει για τι επενδύσει εξαρτώνται από πολλά πράγματα, από συναλλαγματικέ ισοτιμίε, από φορολογικό καθεστώ κτλ. κτλ. Αν θεωρήσουμε ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κρίνουμε αν προσελκύουν περισσότερη ή λιγότερη επένδυση, δεν είμαστε στο σωστό δρόμο. Όταν κανεί επενδύει όμω έχει μια πρόσθετη εξασφάλιση και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην περίπτωση που ανέφερα, Αργεντίνα, η περίπτωση του, της Ιούκος. Μόνο με τη συμφωνία αυτή του ενεργειακού χάρτη μπορούσε κανεί να προσφύγει κατά τον ε, ρωσικού κράτου και να πάρει τα 30 δισεκατομμύρια. Είναι μια ασφαλιστική πολιτική, δεν σημαίνει ότι σε όλες τις περιπτώσεις μπορεί κανείς να είναι σίγουρος. Νομίζω ότι βοηθάει το να πάει κανείς σε μια χώρα και να επενδύσει και γι' αυτό οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται συμφωνίε τέτοιου είδου Τελευταίο σημείο για το θέμα του κόστους ενός διεθνούς δικαστηρίου. Το έχουμε αναφέρει αυτό. Δεν ξέρουμε πόσο θα κοστίσει πραγματικά. Σε ό,τι αποφασίσουμε πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι δευτερεύον θέμα σε σχέση με το αν θέλουμε να το έχουμε αυτό το δικαστήριο ή όχι, γιατί θα φέρει κάποια ε, ωφέλη συγκεκριμένα. Δεν είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά νομίζω πρέπει να το κοιτάξουμε γιατί θα αυξήσει την ασφάλεια δικαίου και θα αφαιρέσει προβλήματα σύγκρουση συμφερόντων όπως αυτά που είπαμε. Κύριε Μπέρτενς δεν θα απαντήσω στα ερωτήματα τα οποία ήδη έχουν τύχει απάντησης. Θα κάνω ό,τι μπορώ για αυτά που αφορούν εμένα. Για, τα, για τη σύγκρουση συμφερόντων των διαιτητών ξέρω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό εν ώψη της κοινή αντίληψης ότι δεν είναι αμερόληπτη. <clears throat> Μπορείτε να κάνετε ένα κατάλογο διαιτητών που τους εμπιστεύεται κανείς ή ένα αρνητικό κατάλογο αυτών που δεν θέλετε. Ίσως θέλετε άτομα που είναι πρώην πολιτικοί, είναι νομομαθείς, είναι καθηγητές δικαίου, αλλά αυτό θα πρέπει να το αποφασίσει κανείς εξ αρχής. Για τα εθνικά δικαστήρια υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά. Θα ήταν καλό τα εθνικά δικαστήρια να αρχίσουν να εφαρμόσουν το διεθνέ δικαίωμα. μέση περιπτώσει δεν έχουν το δικαίωμα να το κάνουμε στο εθνικό σύστημα δικαιοδοσία. Κάποια δικαστήρια το κάνουν, αλλά προτιμούν να μην το κάνουν. Και σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε και ακόμα και στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ισχύει αυτό, για το Policy Space και το άρθρο 20 του GATT έναντι των κανονισμών του ΠΟΕ, πράγματι υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν αιτιολογήσει αυτού του είδου Κάποιε συνθήκε, όχι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά άλλε συνθήκε το κάνουν αυτό. Επομένω, αυτό λειτουργεί με παρά, παρόμοιο τρόπο όπω για τον ΠΟΕ. Γιατί να μην μπορούν να προσφεύγουν οι καταναλωτέ, οι εργαζόμενοι και οι υπέρμαχοι του περιβάλλοντο Εγώ συμφωνώ εδώ. Θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε τέτοιες περιπτώσεις και ενδεχομένω να κάνουν και αυτόνομες προσφυγές. Αλλά το να κάνουν αυτόνομες προσφυγές θα πρέπει να γίνει μέσα σε ένα τελείω διαφορετικό σύστημα. Εγώ προσωπικά το υποστηρίζω, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι πολιτικά εφικτό. Σε ό,τι αφορά την άσκηση πολιτικής πίεσης λόγω της ISDS, Νομίζω ότι πολλές εταιρείες έχουν ήδη προσπαθήσει να ασκήσουν πίεση σε κυβερνήσεις και στο παρελθόν. Αυτό γίνεται πάντα. Πράγματι λοιπόν μπορεί η συμφωνία αυτή να ασκήσει πολιτική πίεση όπως και τα εθνικά και στα εθνικά δικαστήρια μπορούν να είναι ένας τρόπος άσκησης πίεσης. Για τις χώρες που έχουν απομακρυνθεί από αυτό το σύστημα. Η Αυστραλία απομακρύνθηκε αλλά επανέρχεται τώρα και ξαναβάζει το ISDS στις διεθνείς συμφωνίες του. Αυτό έχει να κάνει και με την αλλαγή κυβέρνηση. Επομένω, ίσω και η επόμενη κυβέρνηση να ξανααλλάξει τη γνώμη τη για τι ε, ε, εταιρείε δικηγόρων και τον, το πόσο βγάζουν. Νομίζω ότι βγάζουν γενικά λιγότερο από ό,τι τα μέλη του Κοινοβουλίου. Και για τι εταιρείε οι οποίε βασίζονται σε αυτά τα είδη διατησία, εγώ δεν ξέρω μια εταιρεία νομική μια δικηγορική εταιρεία που ασχολείται μόνο με αυτά τα θέματα. Εγώ δεν ξέρω ποτέ να υπήρξε μια τέτοια εταιρεία. Νομίζω ότι όπως σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ε, νομικών διαμαχών είναι θέμα συμφωνίας με τον πελάτη η αμοιβή του. Και για το αν είναι ε, κομμάτι της συμφωνίας η των ε, μετόχων, πράγματι αυτό πρέπει να γίνει. Και τώρα για τη μεγαλύτερη διαφάνεια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια. Ξέρουμε οι περισσότεροι ποιο είναι το αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να είναι με πιο διαφανής και η διαδικασία. Ο κύριο Ζαν. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, μου έχουν κάνει 7 ερωτήσει. Θα προσπαθήσω βέβαια να είμαι σύντομο. Η πρώτη ερώτηση για το αν η ISDS πρέπει να μπει στο πλαίσιο του ΠΟΕ, αν, αν έχει τη δυνατότητα να διαφυλάσσει το policy space. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι δυνατό στη, διά, στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ε, της συμφωνίας θα πρέπει να μπει στο προήμιο ε, η σχετική αναφορά και επίσης το διατακτικό της συμφωνίας. Αναφορά δηλαδή στην προστασία, ε, δικαιώματα εργαζόμενων, αηφόρα ανάπτυξη, όλα αυτά μπορούν να μπουν στο προήμιο της συμφωνίας μπορούν να μπουν και σε παραπέρα διατάξεις και για μέτρα προφύλαξης για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και αλλού μπορεί να προβλέπονται και γενικές εξαιρέσεις για προστασία ανθρώπινης ζωής, φυτών κτλ. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί τρόποι για να διαφυλαχθεί ο χώρος όπου ασκούν πολιτική τα κράτη και οι σχετικές ρυθμίσεις τους. Δεύτερη ερώτηση. Για ε, συμφωνίες προστασίας ε, επενδύσεων. Πράγματι μας φαίνεται σαν μια πολιτική ασφαλίσεων για τις επενδύσεις και είναι σημαντικό για τις σχέσεις επενδύσεων με χώρες όπου έχουν αδύναμη διακυβέρνηση και όχι μόνο σε ό,τι αφορά την οικονομική νομοθεσία, επενδύσεις κλπ, αλλά και για παράδειγμα ε, στάνταρτ προστασίας των εργαζόμενων κλπ. Εκεί η ε, συμφωνία έχει σημασία για να διασφαλίζει την προστασία των συμφερόντων και των δύο πλευρών. Τρίτη ερώτηση για το regulatory chill, για το ρυθμιστικό πάγωμα δηλαδή, και αν χωρίς το ISDS τι, θα, επιρροή θα έχει στις ροές επενδύσεων. Οι ISDS είναι μηχανισμός επιβολής των προβλεπόμενων της ε, συμφωνίας. Είναι δύσκολο να εξευρεθεί κάποια διασύνδεση, ακόμα και σε μεγαλύτερο πλαίσιο. έχει σχέση με οικονομικές παραμέτρους, πολιτικές παραμέτρους, με, τη, με παραμέτρους διευκόλυνσης των επιχειρήσεων κλπ. Η ερώτηση τώρα γιατί υπάρχει μεγάλη αύξηση διαιτητικών υποθέσεων τα τελευταία χρόνια. Εδώ υπάρχουν διάφοροι παράγοντες. Αφενός η αύξηση επενδύσεων σε αναπτυσσόμενες χώρες, σε φτωχές χώρες δηλαδή, όπως είδαμε πέρσι και πρόπερσι, παραπάνω από ε, τις μισές ροές επενδύσεων πήγανε σε αναπτυσσόμενες χώρες και όπου η διακυβέρνηση είναι ασθενής και εκεί η προστασία των επενδυτών είναι ασθενής και γι' αυτό το 70% των υποθέσεων διακόπτει ο πρόεδρος. Εδώ πρέπει να σας διακόψω ε, κύριε Ζαν. Κύριε Χίντελανγκ. Άλλες τρεις ερωτήσεις έπρεπε να απαντήσω. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Ε, πώς να αποφύγουμε την ε, αντίληψη περί των διεθνών επενδυτικών ε, συμφωνιών το καλύτερο θα ήταν να έχουμε ένα μόνιμο δικαστήριο με δικαστές ε, αλλά αν αυτό δεν είναι εφικτό από πολιτικής άποψης, τότε ίσως θα μπορούσε κανείς να... αλλάξει την αντίληψη, δηλαδή να υπάρχει περισσότερη διαιτησία από ότι τους διαιτητές που αυτή τη στιγμή δρούν σε αυτό το πεδίο. Γιατί κάθε ένας τότε θα ωφελούταν λιγότερο από κάθε απόφαση. Όσον αφορά το θέμα της, της ε, νοσιακής νομοθεσίας, της ΕΤΑ και άλλων ε, μεχανισμών επίλυσης διαφορών της Ένωσης, θα πω το εξής. Το δικαστήριο είναι ιδιαίτερα ε, εγωιστικό και δηλότυπο ε, όσον αφορά το δικό του μονοπόλιο ερμηνείας ε, και του, του, της κοινοτικής νομοθεσίας, δηλαδή το απόλυτο δικαστήριο, και ε, ε, και κρίνει κατά πόσο η διαιτησία του κράτους μέλους επηρεάζει το κοινοτικό δίκαιο και άρα το δικαστήριο εκεί πρέπει να αποφασίσει εάν και κατά πόσο αρκεί αυτός ο αντίκτυπος για να κινητοποιηθεί και να ισχύσει το κοινοτικό δίκαιο αλλά η γνωμοδότηση 213 και 109 σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα προς τα εκεί κλείνουν Υπάρχει και το θέμα της τρέβλεσης των αρμοδιοτήτων για το ΔΕΚ. Ελπίζουμε πως ε, ένας μηχανισμός που προβλέπει η Κομισιόν για να καθορίζει το σωστό αποδέκτη ε, είναι συμπαγής, είναι ε, σταθερή και σε σχέση με τα εθνικά συστήματα και το STS, εγώ προσπάθησα αυτό να το τοποθετήσω, ε, να το δώσω με την εικόνα ενός ε, ε, κρουαζιερόπλιου και, ενός, και μια σωστική λέμβου. Αυτό που θα μπορούσε να είναι δηλαδή το γερμανικό ή το βρετανικό ή το γαλλικό σύστημα, δηλαδή έχει βρεθεί και μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στο ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αναγνωρίζεται από τον πληθυσμό, θεωρείται δίκαιο εν γέννη το σύστημα αυτό και στα ανεπτυγμένα νομικά συστήματα εν γέννη αποδεχόμαστε τις αποφάσεις των διεθνών δικαστήριων εάν το Εθνικό Δικαστήριο θεωρηθεί ότι έχει υπάρξει ότι έχει κάνει διακριτική μεταχείριση όπως δείχνει συνήθως το, το δικαστήριο θα πίνει δικαιωμάτων. Σας Πάμε στο δεύτερο μέρος της ακροάσεως. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε λοιπόν στο δεύτερο τμήμα της ε, για τις ρυθμιστικές πτυχές του, της συμφωνίας TTIP. Όπως είπα, είναι και συνέχιση της ακρόασης που κάναμε το Φεβρουάριο πέρσι με τίτλο «Συνεκτικότητα στο ρυθμιστικό επίπεδο και εφαρμογή των κανόνων στο πλαίσιο του TTIP». Τότε δεν ξέραμε σχεδόν τίποτα για το, την εμβέλεια και το περιεχόμενο του αντίστοιχου κεφαλαίου για την TTIP. Αυτή τη φορά ξέρουμε περισσότερο. Προχωρούμε προς μια κομβική στιγμή στις διαπραγματεύσεις, γιατί ο 8ος γύρος των διαπραγματεύσεων TTIP την επόμενη εβδομάδα θα εστιάσει πάρα πολύ στις ρυθμιστικές πτυχές. Η Κομισιόν ετοιμάζουν τώρα την ε, πρακτική δράση και τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν σε ό,τι αφορά την ευρωστία σε επίπεδο ρύθμισης, την ευφυά ρύθμιση, την ε, κατευθυνόμενη από πολιτική κατεύθυνση ρύθμιση, τη διαβούλευση με εμπλεκομένους δευτερεύουσες ε, ενέργειες, μείωση του διοικητικού άχθους. Όλες αυτές οι πτυχές λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικές και υπογραμμίζονται και από την Αμερικανική πλευρά στις διαπραγματεύσεις. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα από την Κομισιόν και μετά από δύο ακαδημαϊκούς ένας από τους οποίους είχε ήδη παραστεί ενώπιόν μας το Φεβρουάριο, ο κύριος Αλεμάνο. Καλώς ήλθατε λοιπόν και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίσης έχουμε ένα εκπρόσωπο από την Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία σε ό,τι αφορά το χρόνο. Μέχρι τώρα ο κύριος Αλεμάνο θα πρέπει να έχει τελειώσει την ομιλία του. Ο μάλλον συγγνώμη, ο κύριο Πεχόντε Πνίνκα θα είχε μιλήσει 10 λεπτά και ο κύριος Αλμάνο θα ήταν στη μέση της ομιλίας του. Σας παρακαλώ λοιπόν, μήπω δεν μπορεί, μήπως θα μπορούσατε να μην χρησιμοποιήσετε πλήρω τα 15 σας λεπτά διακεκριμένη καλεσμένους μας για να μείνει και λίγος χρόνος για ερωτήσεις και απαντήσεις μετά από την έγκριτη παρέμβασή σας. Ο πρώτος ομιλητής λοιπόν είναι ο κ. Φέρνατο Περροντεπινίνκα από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το λόγο έχετε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου προσφέρετε την ευκαιρία να σας εξηγήσω πού βρισκόμαστε για τα αριθμιστικά θέματα της συμφωνίας TTIP να σας εξηγήσω τι συζητούμε, ποια ρυθμιστικά θέματα τίθενται και ποια δεν τίθενται και να σας αναπτύξω και ορισμένα στοιχεία για τους βασικούς πυλώνες της συζητήσεως και να καταλήξω και στο λεγόμενο state of play, δηλαδή που βρισκόμαστε. Και πρώτα υπενθυμίζω την εντολή που μας κατευθύνει στο έργο μας. Για ρυθμιστικά θέματα η συμφωνία έχει το στόχο να αφαιρέσει περί τους φραγμούς για τις επενδύσεις μεταξύ αυτών και μη εμπορικούς φραγμούς, non-trade buyers, να φτάσει σε ένα φιλόδοξο επίπεδο ρυθμιστικής ε, συμβατότητας, αμοιβαίας αναγνώρισης, εναρμόνισης και βεβαίως χωρίς να θίξει το δικαίωμα των μερών να ε, ε, ρυθμίζουν στο επίπεδο που θεωρούν κατάλληλο. Εδώ λοιπόν η λέξη κλειδί είναι περιττή φραγμή. Η εντολή στις διαπραγματεύσεις για τις οποίες συζητούμε χωρίζεται σε τομείς φυτικά και φυτογειονομικά μέτρα, SPS. Δεν θα έρθω σε αυτά τόσο πολύ τώρα. Στα τρία άλλα περισσότερο. Τεχνική φραγμή στο εμπόριο. Για παράδειγμα διαδικασίες ε, εναρμόνισης, τεχνικές απαιτήσεις, οτιδήποτε δηλαδή ρυθμίζει το εάν κάποιο προϊόν μπορεί να διατεθεί στο εμπόριο στην επικράτεια μιας χώρας. Η νομοθετική συνοχή γενικότερα που προβλέπει γενικότερες κατευθύνσεις διατομιακές που επιτρέπουν την άσκηση ρυθμιστικών πρακτικών με στόχο την βελτίωση της συνοχής ή την αποφυγή ασυμβατοτήτων που είναι περιττές μεταξύ πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, τομεακές διατάξεις, ειδικέ ρυθμίσεις δηλαδή για ειδικού τομείς που θα ε, συναποφασιστούν. Ορισμένες τώρα βασικές έννοιες που διέπουν το έργο μας. Τι σημαίνει ρυθμιστική συνοχή. Όπως είπα, η μείωση περιττών ρυθμιστικών ασυμβατοτήτων, κατάργηση επικαλύψεως διαδικασιών που δεν είναι απαραίτητες, ασυνεπών απαιτήσεων προϊόντων, διπλών δοκιμών και ούτω καθεξής. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Το γεγονό δηλαδή ότι και οι δύο πλευρέ έχουν αναπτύξει ρυθμίσει, τεχνικέ ρυθμίσει κτλ. χωρί να εξετάζουν ποια είναι η εμπειρία τη άλλη πλευρά. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι έχει έρθει η ώρα τώρα να εξετάσουμε λίγο τι ρυθμίσει μα να δούμε πώ μπορούμε να τι βελτιώσουμε σε κοινή προσπάθεια, να δούμε δηλαδή πού μπορούμε να εξορθολογήσουμε τι προσπάθειές μα, όπου οι ρυθμίσεις μας είναι είτε συγκρίσιμες είτε ισοδύναμες. Για παράδειγμα, έχουμε ένα είδος εργαλειοθήκης. Αμοιβαία αναγνώριση ρυθμισών εφόσον υπάρχει βέβαια ισοδυναμία. Κάποια εναρμόνιση ή ευθυγράμμιση απαιτήσεων σε ορισμένες περιπτώσεις η θέσπιση κανόνων που θα ισχύουν και στις δύο πλευρές η εφαρμογή κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, η εφαρμογή δηλαδή διεθνών κανόνων ή προδιαγραφών. Η μέθοδος για να επιτευχθεί αυτό είναι συνεργασία μεταξύ ρυθμιστών των δύο πλευρών. Δεν είναι πολιτική διαδικασία αυτή, το τονίζω. Είναι διαδικασία όπου οι ρυθμιστές θα πρέπει να δηλώσουν ικανοποιημένοι ότι μπορεί να υπάρξει εξορθολογισμός των όσων πράττουν και οι δύο πλευρές στη βάση τεχνικών αξιολογήσεων των δεδομένων. να σας δείξω τρεις διαφάνειες σχετικά με το τι δεν σημαίνει ε, ρυθμιστική ε, συνοχή. Άρα δεν σημαίνει μια διευρυμένη, μια γενικευμένη αμοιβαία αναγνώριση και εναρμόνιση. Δεν μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν ρεαλιστικό ούτε τεχνικά ούτε και πολιτικά. Δεν θα υπάρξει κοινή νομοθεσία, δεν θα υπάρξει κάποιο κοινό όργανο που θα έχει την ικανότητα να εκδίδει ε, ρυθμίσεις δεν θα υπάρχει επηρεασμό της ρυθμιστικής κυριαρχίας οποιασδήποτε των πλευρών αυτό θα το προτείνουμε εμείς τουλάχιστον πολύ ξεκάθαρα δεν υπάρχει δηλαδή υποχρέωση να προκύψουν αποτελέσματα από τη συνεργασία δεν θα υπάρχει διαπραγμάτευση για στόχους και επίπεδα ε, προστασίας καμία από τις, από τις ε, πλευρές δεν θα πρέπει να προσπαθήσει να επιβάλλει αλλαγή τρόπου ρυθμίσεως, γιατί βεβαίω και οι δύο πλευρές θα αντισταθούν λυσασμένα, ούτε θα επιτραπεί η TTIP να επιβραδύνει την νομοθετική διαδικασία. Επίσης η περίφημη ρυθμιστική συνοχή δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει η ισορροπία της εκπροσώπησης των ενδιαφερομένων, stakeholder δηλαδή. Όλοι θα πρέπει να την χάνουν ισοδύναμης, ισότιμης μάλλον μεταχείρισης στην πράξη. Είτε δίνοντας την άλλη πλευρά την δυνατότητα, την ικανότητα να επηρεάσει τη ρυθμιστική ε, μας ε, διαδικασία. Δεν πρόκειται να προσφέρουμε μια 21 η θέση στο Συμβούλιο Υπουργών για τους Αμερικανούς, ούτε και ανάποδα βεβαίως έτσι, ούτε πρόκειται να δημιουργήσουμε μια διατλαντική ενιαία αγορά που οι κανόνες της να υπηρεσίουν των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς. Έτσι συνοψίζοντας, η ρυθμιστική συνοχή δεν σημαίνει ότι παρετείται κανείς ή μειώνει την ε, προστασία που εγγυώνται οι συνθήκες και οι νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι ούτε τεχνικά ούτε νομικά δυνατό ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στις ΗΠΑ. Έχουμε περάσει τώρα πλέον νομίζω 300 ώρες γύρων διαπραγματεύσεων και δεν έχω ακούσει σε καμία περίπτωση κανένα ρυθμιστή να προτείνει οτιδήποτε το οποίο θα σήμαινε μείωση του επίπεδου προστασίας. Δεν έχω λοιπόν κανένα λόγο να σκεφτώ ότι αργότερα θα προκύψουν τέτοιες προτάσεις. Για την ώρα πάντως δεν έχουμε δει οποιαδήποτε τέτοια πρόταση, ούτε προφορικά ούτε γραπτός. Και η δέσμευσή μας είναι να προστατεύσουμε τον τρόπο με τον οποίο ε, θεσπίζουμε τις νομοθετικές μας ρυθμίσεις. Εκεί που θέλουμε να δώσουμε προσοχή είναι στους τομείς εκείνους όπου μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα και να εισαγάγουμε ε, νομοθετικά μέτρα που να μειώσουν το κόστος. Στο κεφάλαιο τώρα για την ε, ρυθμιστική συνοχή, εκεί θα προβλέπονται ορθές ρυθμιστικές πρακτικές, διαφάνεια, έγκαιρη προειδοποίηση, διαβούλευση των, με τους ε, ενδιαφερομένους, ε, μελέτες αντικτύπου, ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των ρυθμιστών, ώστε και οι δύο πλευρές να γνωρίζουν ποια πράγματα επίκυνται να προταθούν, είναι στον αγωγό όπως λένε, και να μπορούν να γνωρίζουν τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της η άλλη πλευρά και να μπορούν να αναζητήσουν λύσεις κοινά εποφελής για καλύτερη νομοθετική ρύθμιση, χρησιμοποιώντας διάφορα μέτρα, αναμοιβή αναγνώριση, απλούστευση, απλοποίηση σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Θα αρχίσουμε βεβαίω να συζητούμε πρώτα από αυτούς, όχι για τομείς όπου έχουμε τελείως διαφορετική προσέγγιση στην προστασία του κοινού συμφέροντος δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε μονάχα τη μείωση του κόστους με το διατλαντικό εμπόριο θα προωθήσουμε την ρυθμιστική συνοχή και παγκοσμίω. Οι σχετικές αυτές βασικές αρχές θα πρέπει να διατηρηθούν μεταξύ αυτών και η αρχή της προφύλαξης precautionary principle δεν πρόκειται να ζητήσουμε από τις ΗΠΑ να δεχτούν την αρχή προφύλαξης. Το βασικό στοιχείο είναι ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να σέβονται το ρυθμιστικό σύστημα της άλλης πλευράς. Τώρα τελικοποιείται το κείμενο για το όργανο ρυθμιστικής συνεργασίας και ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα μπορέσει να δημοσιευτεί. Δύο λόγια για το όργανο τώρα της ρυθμιστικής συνεργασίας που θα έχει το σκοπό να παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμιστικών διατάξεων της TTIP. Δεν θα έχει όμως εξουσίες νομοθετικές. Ούτε θα έχει και την αρμοδιότητα να αξιολογεί τα σχέδια των ρυθμίσεων της άλλης πλευράς. Δεν θα καθυστερεί έτσι επομένως την ε, υιοθέτηση των σχετικών ρυθμίσεων. Ούτε θα προσφέρει τη δυνατότητα στην άλλη πλευρά να επηρεάζει ρυθμιστικές αποφάσεις. Και βεβαίω θα πρέπει να διεξάγει το έργο του με διαφάνεια, με υποβολή αναφορών και με το σχετική παρακολούθηση, monitoring. Ο στόχος είναι η επίτευξη συγκεκριμένων απτών αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Μιλούμε για όλους τους τομείς όπως των αυτοκινήτων οχημάτων, τεχνολογίας, χημικών, ζυζανιοκτώνων, υφαντουργικό τομέα. Είναι βέβαια νωρίς να πει κανείς που θα καταλήξουμε ακόμα ποια είναι η έκβαση, όμως υπάρχει υψηλό επίπεδο κοινού ενδιαφέροντος. Με λίγα παραδείγματα τώρα που φαντάζομαι θα τα συζητήσει και ο Ζόναρτ, τα αυτοκίνητα οχήματα. Εκεί επιθυμούμε να επιτύχουμε αμοιβαία αναγνώριση ισοδυναμίας από όσο δυνατό περισσότερο τεχνικών ρυθμίσεων και στη βάση ε, τεχνικών αξιολογήσεων. Στα χημικά τώρα για παράδειγμα έχουμε πολύ διαφορετικά συστήματα. Δεν υπάρχει τρόπος λοιπόν να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση. Αντίθετα εκεί ρίχνουμε ε, την προσπάθειά μας σε μια συνεργασία ανάπτυξης κοινή μεθοδολογίας για να αποφύγουμε οποιασδήποτε περιττές επικαλύψεις και βέβαια και με σεβασμό του χρονοδιαγράμματος και των προθεσμιών που επιβάλλουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις και των δύο πλευρών. Τέλος, το που βρισκόμαστε, state of play. Ακόμα είναι κάπως νωρίς να πει κανείς τι ακριβώς θα συμφωνηθεί. Προφανώς. η προέλευσή μας είναι πολύ διαφορετική σε ό,τι αφορά τη ρυθμιστική συνοχή. Δηλαδή ερχόμαστε από τελείως διαφορετικές πλευρές. Αλλά υπάρχει τόπος συνεργασίας. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι θα συνεχίσουμε να επιζητούμε μια ανοιχτή διαφανή διαδικασία για να μπορεί το κοινό να παρακολουθεί περί τίνος πρόκειται. Το συμπέρασμα εν τέλει είναι ότι έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας έχουν γίνει πολλά πράγματα για να διευκρινιστεί το τοπίο, να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Χρειάζεται όμως ακόμα πολύ δημόσια συζήτηση, όπου ευχαρίστω θα την διεξαγάγουμε μαζί σας. Thank Σας ευχαριστώ που μας ε, εξοικονομήσατε λίγο χρόνο για ερωτήσεις αλλά και απαντήσεις. Ο καθηγητής Αλεμάνο, καθηγητής Ζωάν Μονέ για τον Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και την έρθμιση του κινδύνου έχει το λόγο ο κ. Αλεμάνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε πρωτού ξεκινήσω, θέλω να αναφέρω μια επιφύλαξη. Είναι αυτά που θα σας πω συμπέρασμα μιας έκθεσης πολιτικής που είχα προετοιμάσει το 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι είχε συζητηθεί από την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Όπως ακούσαμε και στην προηγούμενη παρουσίαση και πώς το ξέρουμε όλοι και γι' αυτό γίνεται αυτή η ακρόαση σήμερα, οι διαπραγματεύσεις TTIP ήταν ιδιαίτερα αμφιλεγόμενες και ιδίω σαν εμπορική συμφωνία υπάρχουν πολλές αποχρώσεις τα, δεν εμπλέκονται πάντα τα ίδια κράτη-μέλη αλλά υπάρχουν τρία βασικά θέματα που μονοπολούν την ε, προσέγγιση της κοινή γνώμης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πρώτο θέμα είναι το θέμα της διαφάνειας. Το δεύτερο είναι ισοπαίδωση προς τα κάτω που αντιμετωπίστηκε εν μέρει από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν και το τρίτο ήταν το θέμα του ISDS που αναφέρθηκε στο προηγούμενο πάνελ. Το πρώτο που θα ήθελα εγώ να πω είναι ότι υπάρχουν περαιτέρω θέματα πέραν αυτών των τριών στην TTIP. Υπάρχει το θέμα του πολιτικού και δημοκρατικού ελέγχου τη συμφωνίας αυτής, η οποία είναι υποδιαπραγμάτευση, αλλά και από τη στιγμή που θα τεθεί σε εφαρμογή αυτή η συμφωνία υπάρχει το θέμα της εφαρμογής που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τι θα γίνει εάν υπάρξει έγκριση αυτής της συμφωνίας. Ένα άλλο σημείο είναι το θέμα της ισορροπίας των δεσμεύσεων μεταξύ των δύο συμβαλόμενων μερών. Αν σας ρωτήσω τι είναι το TTIP, πιστεύω ότι κάποιοι οι οποίοι είναι υπέρμαχοι θα πούν ότι είναι μια συμφωνία εμπορικού χαρακτήρα νέας γενιάς. Αν ακούσουμε την άλλη πλευρά θα πούν ότι είναι περισσότερο ένα διεθνέ ρυθμιστικό πλαίσιο. Δημιουργούμε ένα νέο είδος διακυβέρνηση μεταξύ ομογενών ή ομοιογενών καλύτερα ε, φορέων όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ηνωμένη Ευρώπη. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν γιατί θέλουμε μια τέτοια συμφωνία και πώς θα την κάνουμε αυτή τη συμφωνία. Οι λόγοι για τους οποίους έχουμε αυτή τη διαπραγμάτευση είναι για να ξεπεράσουμε τους λεγόμενους φραγμούς πίσω από τα σύνορα που έχουν αναφερθεί εδώ και πολλά χρόνια ως μη τελωνιακή φραγμή και είναι ουσιαστικά το θέμα των εθνικών ρυθμίσεων. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Η TTIP δεν είναι σε κενό αέρος, ξέρουμε ότι βασίζεται στο καθεστώς του ΠΟΕ, για αυτό το λόγο πόσες φορές έχουν αναφερθεί αυτές οι συμφωνίες και επίσης βασίζεται στην ρυθμιστική συνεργασία διατλαντικού χαρακτήρα που εδώ και χρόνια και δεκαετίες λαμβάνει η χώρα. Υπάρχει λοιπόν διάλογος και υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες στο τομεακό επίπεδο, όπως χάρη η αναγνώριση αμοιβαίων ε, συμφωνιών όπως αυτή για τα βιολογικά προϊόντα. Ο ΠΟΕ έχει δώσει μια κοινή προσέγγιση το 1995 λέγον ότι με το να περιοριστεί η δυνατότητα των ε, μελών να δράσουν θα πρέπει να ακολουθηθεί μια σαφής κατευθυντήρια γραμμή για τους τεχνικούς φραγμούς που δεν είναι αυτοί που αφορούν τη δημόσια υγεία, SPS. Πρόκειται λοιπόν για εναρμόνιση που εμποδίζει, περιορίζει την δυνατότητα των κρατών μελών για να ρυθμίσουν, γιατί λένε ότι πρέπει να μήπως μπορείτε να πατήσετε λίγο φρένο διότι οι διερμηνείς δεν σας προφέρουν, λέει ο πρόεδρος. Βλέπουμε λοιπόν την εμπειρία του ΠΟΕ και είναι σαφές ότι η εμπειρία αυτή δεν επαρκεί. Εκεί ακριβώς είναι η αλλαγή στην οτροπία της TTIP. Ας δούμε λοιπόν πώς αναπτύσσεται αυτή η σχεδίαση της TTIP. Η TTIP προσπαθεί να προχωρήσει λίγο περισσότερο στην προσπάθεια του συντονισμού το, της του εμπορίου. Αν δείτε σε τι συνίσταται και οι ιδέες την διατρέχουνε, στις διαπραγματεύσεις υπάρχει αυτή η ιδέα ότι η συνεργασία εστιάζεται για το πώς ρυθμίσουμε και όχι το τι ρυθμίσουμε και ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να υπάρξει σύγκληση σε ενιαίες διαδικασίες. Αν λοιπόν ακολουθήσουμε παρόμοιες διαδικασίες είναι η ιδέα, έχουμε περισσότερες πιθανότητες να φτάσουμε σε κοινά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να βοηθήσουμε να υπάρξει μια ουσιαστική σύγκληση. Έχουμε το παράδειγμα τη συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά που δεν είναι εμπορική συμφωνία αλλά είναι μια μορφή διεθνού, ρυθμιστικής συνεργασίας αλλά και συμφωνία ΣΥΤΑ η οποία έχει προαναφερθεί. Αν περάσουμε και πέραν τη ΣΥΤΑ η TTIP θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα μόνιμο τρόπο συνεργασίας σε ρυθμιστικό επίπεδο που μπορεί να ξεπεράσει και το κλίμα διαπραγματεύσεων το οποίο διέπει τις περισσότερες εμπορικές συμφωνίες και ενδεχομένω να ξεπεράσει διαφορές οι οποίες είναι ιδεολογικού χαρακτήρα μέσω μιας ζωντανής συμφωνίας. Μια συμφωνία η οποία μπορεί να εμπλουτίζεται συνέχεια με συμφωνίες. Αυτό το οποίο δείχνω στους φοιτητέ μου και εσείς ξέρετε περισσότερα από τους φοιτητέ μου για να καταλάβετε τι γίνεται στην TTIP αλλά θέλω να σας δείξω αυτή τη διαφάνεια. Πρόκειται για το εξή παιχνίδι να συμφωνήσουμε σε μια οριζόντια ε, διαδικασία, μια οριζόντια πειθαρχία που θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για να συμφωνούν οι ρυθμιστέ σε συγκεκριμένου τομεί, αλλά συγχρόνω να μπορέσουμε να επιτύχουμε και μια τομεακή κάθετη προσέγγιση. Ορισμένε συμφωνίε λοιπόν θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό είναι λοιπόν ένα δύσκολο παιχνίδι για να παίξει κανεί, γιατί και οι δύο πλευρέ θα πρέπει να <clears throat> υποστηρίξουν και τις δύο προσεγγίσεις. Από τη μία πλευρά λοιπόν έχουμε ένα κεφάλαιο οριζόντιας ρύθμισης και από την άλλη μεριά έχουμε ένα κάθετο τομεακό κεφάλαιο. Αν δούμε λοιπόν την εμβέλεια αυτή τη συμφωνία, όπω είπε και πρόσωπο τη Κομισιόν, όλα τα μεταγενικέ εφαρμογέ που έχουν κάποια διατλαντική διάσταση θα πρέπει να υπόκεινται στην πειθαρχία τη ΤΤΙΠ. Το θέμα είναι ποια είναι αυτά τα θέματα και εδώ θα πρέπει να είμαστε λίγο επιστημονικότεροι αλλά ένεκα της φύσης των νομοθετικών πράξεων στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη μπορούμε να πούμε εν γέννη ότι περισσότερο από αυτούς τους κανόνες στις ΗΠΑ είναι μη νομοθετικές πράξεις που είναι εκτελεστικού χαρακτήρα ε, νόμων του Κογκρέσου των ΗΠΑ, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι νομοθετικού χαρακτήρα κατά πάσα πιθανότητα αν δούμε την οριζόντια πειθαρχία. Είναι τέσσερα κυρία καθήκοντα τα οποία επιβάλλονται και στι δύο πλευρέ του Ατλαντικού για να υπάρξει αυτό το μόνιμο φόρουμ, να υπάρξει ένα μηχανισμό έγκαιρη προειδοποίηση, να εξασφαλίσουμε το διάλογο και ενδεχομένω να έχουμε και μια αξιολόγηση αντικτύπου για να δούμε την, τον αντίκτυπο για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αν δούμε του μηχανικού, του μηχανισμού, μάλλον, όχι του μηχανικού, και προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε στις πραγματικότητες. Εδώ θα έπρεπε να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ της εφαρμογής αυτής της ε, πειθαρχίας σε νέους κανονισμούς, σε μη υπάρχοντες κανονισμούς, οι οποίοι μπορεί να έλθουν στο μέλλον γιατί αντιμετωπίζουν παραγωγικά τεχνολογικές εξελίξεις όπως οι νανοεφαρμογές και υπάρχοντες κανονισμούς, υπάρχοντες ρυθμίσεις. Μία από τις επιλογές λοιπόν που έχει αναφερθεί στην βιβλιογραφία και από τους ε, ε, λήπτες αποφάσεων και πάλι σας παρακαλώ να είσαστε πιο βραδείς. Οι μηχανισμοί οι οποίοι φαίνεται να αποκρίνονται αυτή τη στιγμή είναι η αξιολόγηση ρυθμιστικής συμβατότητας. Η ιδέα του να φτιάξουμε λοιπόν μια στην μια επαφή μεταξύ ρυθμιστών που θα αρχίσουν να αναρωτιόνται για το πρόβλημα αυτό. Θα πούνε έχουμε το ίδιο πρόβλημα όταν αντιμετωπίσουμε μια συγκεκριμένη τεχνολογία και συνέχεια να προσπαθήσουν να βρουν αποτελέσματα ή αναλυτικέ μελέτε οι οποίε μπορούν να είναι αμοιβαία συνεκρίσιμε και επίση να αναλύσουν ποιο είναι το κόστο αν ακολουθούμε διαφορετικέ λύσει για τα προβλήματα. Αν δούμε λοιπόν αυτέ τι λύσει για του κανονισμού που υπάρχουν θα λειτουργεί διαφορετικά θα είναι πιο κοινού χαρακτήρα γιατί έχουμε τόσο πολλού κανονισμού και από τι δύο πλευρέ του Ατλαντικού. Η διαδικασία θα ξεκινούσε όπω και στην περίπτωση Καναδά Ηνωμένων Πολιτειών με ένα σύστημα αναφορών όπου οι εμπλεκόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τι ρυθμίσει να κάτσουν γύρω από το τετράγωνο τραπέζι και να δουν τα στοιχεία σε σχέση με τα ισοδύναμα αυτών των προτύπων και να μπορέσει να προκύψει λοιπόν μια διαβούλευση, ενδεχομένω μια δημόσια κρόαση. Ακούσατε για πολλά παραδείγματα θα δείτε τα παράδειγματα σε λίγο από την αυτοκινητοβιομηχανία που, είναι, ε, που εξηγούν τα μόνα τους την πραγματικότητα. Αλλά υπάρχει μια γενική ανησυχία που πρέπει να λάβουμε όλοι υπόψη κατά πόσο αυτός ο μηχανισμός θα οδηγήσει σε ισοπαίδωση προς τα κάτω. Δηλαδή, επειδή και μόνο υπάρχει αυτός ο μηχανισμός, δημιουργούμε κίνητα και για τους ρυθμιστές από τις δύο πλευρές να μειώσουν τα πρότυπά τους. Κατά την άποψή μου και επί τη βάση που σας περιέγραψα προηγουμένως, η απάντηση θα πρέπει να είναι νιέτ η αυτονομία στο ρυθμιστικό τομέα θα πρέπει να διατηρηθεί, οι πλευρές οι οποίες κάθονται στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων θα δεσμεύονται από συμφωνία μόνο αν υπάρξει μια συμφωνία. Απουσία τέτοια συμφωνίας θα παραμένει απλώς αυτό το οποίο υπάρχουν όμως και πολλά ανοιχτά ερωτήματα, κάποια έχουν αντιμετωπιστεί, κάποια ανοίγουν τώρα. Θα πρέπει να δούμε και τι θα γίνει μετά από την σύναψη μια συμφωνία, εάν τύχει έγκριση σε αυτή η συμφωνία, πώ θα εφαρμόσουμε λοιπόν αυτό το κεφάλαιο, ποιο θα το εφαρμόσει, τι θα συμβεί από τη στιγμή που ένα κεφάλαιο θα τεθεί σε λειτουργία. Και εδώ προτείνω να κάνουμε διάκριση μεταξύ δύο χρονικών στιγμών. Την στιγμή τη εφαρμογή αυτή τη πειθαρχία και τη στιγμή τη μεταγραφή. Πρώτα απ' όλα, πώ θα μπορέσουμε σε θεσμικό επίπεδο, σε επίπεδο θεσμική σχεδίαση να λειτουργήσουμε το διάλογο αυτό μεταξύ ρυθμιστών στην Ευρώπη και στι Ηνωμένες Πολιτείες και μόλις μπορέσει να επιτευχθεί σε ένα συγκεκριμένο τομέα μια συμφωνία, παραδείγματο χάρη για τα αυτοκίνητα, πώς κάθε πλευρά θα εφαρμόσει αυτή τη συμφωνία στο δικό τη σύστημα. Και το μεγάλο ερώτημα, το οποίο σα ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι ποιο θα είναι ο ρόλο των συνομοθετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα κληθούν να παίξουν σε αυτή τη διαδικασία και ιδίω ποια θα είναι και η συμμετοχή του κοινού. Ένα από τα μοντέλα τα οποία έχουν παρουσιαστεί στην θεσμική σχεδίαση είναι το Συμβούλιο Ρυθμιστικής Συνεργασίας, το οποίο θα κάνει αυτήν την άσκηση βασιζόμενο σε επιτροπές ανάτομης. Και το ερώτημά μου είναι ποιος θα κάθεται σε αυτές τις επιτροπές, οι ρυθμιστές, οι αρμόδιοι για το εμπόριο και πώς όλα αυτά εξασφαλίζουν τη θεσμική ισορροπία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τώρα έρχεται το κύριο μήνυμα το οποίο ήθελα να σας δώσω όταν ισχυρίστηκα ότι το κύριο θέμα για την TTIP δεν θα είναι, δεν θα πρέπει να είναι αυτό που συζητούν σήμερα τα μέσα ενημέρωση, αλλά ένα πιο λεπτό σημείο που θέλω να αναφέρω. Το TTIP θα γίνει ένας καινοτόμος μηχανισμός διακυβέρνησης ο οποίος θα προσπαθήσει αδειρήτως να ξανανοίξει τη διαδικασία ρυθμίσης και νομοθεσίας, όπου εξασφαλίζεται η ισοδυναμία δύο συστημάτων θα πρέπει να ξανανοίξει η νομοθετική διαδικασία. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει κάποια συμμετοχή στη διαδικασία αυτή και κάποιος πολιτικό έλεγχος για τη φάση της εφαρμογής της συμφωνίας. Για να σας δώσω άλλη μία εικόνα, υπάρχει μία ένταση μεταξύ της ανάγκης για αποτελεσματικότητα για να λειτουργήσει η συμφωνία, αλλά από την άλλη μεριά χρειάζεται και πολιτικός έλεγχος. Εν κατακήρυ, το TTIP από μόνο του δεν θα μειώσει την αυτονομία των ρυθμιστών για τις δύο πλευρές των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής, αλλά και θα διατηρήσουν την αρμοδιότητα οι δύο πλευρές για να αποφασίσουν αν θα έχουν νέου κανόνες ή να αναγνωρίσουν ως ισοδύναμους κανόνες που υπάρχουν, αλλά αναπόφευκτα η φύση, το σχήμα και ο βαθμός αυτής της ρυθμιστικής συνεργασίας μπορεί να χρειαστεί εξισορρόπηση μεταξύ δημοκρατικού ελέγχου και αποτελεσματικότητας. Όταν σκεφτόμαστε λοιπόν για το οριζόντιο κεφάλαιο του TTIP, σκεφτείτε για τη γέφυρα που θα μπορέσουμε να φτιάξουμε, η οποία θα συνδέει τις δύο, τις δύο όχθες του Ατλαντικού, επί τη οποία γέφυρα μπορεί να πηδήσουν οι ρυθμιστέ, αλλά κανείς άλλος δεν θέλει ενδεχομένω να χρησιμοποιήσει αυτή τη γέφυρα. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Or Goes to Professor uh, Fizan, Professor in Public Law and Theory of Law of Και τώρα έχουμε τον ε, κύριο Φραν. Ευχαριστώ μου ε, περιποιεί μεγάλη τιμή το γεγονό που την προσκαλέσατε. Θα αναφερθώ ναι, σε τέσσερα ε, θέματα. Δύο περί δημοκρατίας και δύο περί περιεχομένου των προδιαγραφών. Πρώτο, σύντομο. Αυτό αυτός είναι που δεν έχει. Οι δημοκρατικοί στις ΗΠΑ προσπαθούν να επιβάλλουν und να επιβάλλουν η απόφαση για την TTIP αλλά και για την ΣΕΤΑ να περιλαμβάνει και επιμέρους διορθώσεις, δηλαδή το Κοινοβούλιο να μπορεί να αποφασίζει για εξαιρέσεις και άλλες λεπτομέρειες. Αυτό είναι ασύνηθες στις διεθνείς συμβάσεις. Ως Κοινοβούλιο δηλαδή λαμβάνετε το κείμενο και σας λένε ή σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Δεν μπορεί κανείς να δεν μπορεί ένα κοινοβούλιο να επιφέρει βελτιώσει ή διορθώσει. Αυτό λοιπόν το μοντέλο προτείνουν οι δημοκρατικοί στι ΗΠΑ μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Δεύτερο, όταν μιλούμε για την ρυθμιστική αρχή και τη μελλοντική ρυθμιστική αρχή τη TTIP, δεν μπορούμε και πολλά πράγματα γιατί δεν υπάρχουν ακόμα τα κείμενα. Μπορεί να δει κανεί ποια είναι τα αποτελέσματα τη διαπραγμάτευση στην ΣΕΤΑ. Και τα κοίταξα εγώ προσεκτικά. Στη διαπραγμάτευση λοιπόν τη ΣΕΤΑ, ε, τα είδατε αυτά και σε κάποια διαφάνεια πριν, σε διάφορους τομείς προβλέπονται εξειδικευμένες επιτροπές που είναι αρμόδιες για τελωνιακά, για προστασία περιβάλλοντος και ούτε καθεξής. Αυτές οι επιτροπές παράγουν έργο που πηγαίνει σε μια κοινή επιτροπή, joint committee, και κάνουν προτάσεις για ρυθμίσεις ανατομέα. Στο δικό του λοιπόν τομέα αρμοδιότητας. Έρχεται τώρα το κρίσιμο θέμα γιατί αυτή η κοινή επιτροπή, η Joint Committee, θα λαμβάνει δεσμευτικές για τα μέρη αποφάσεις για ορισμένου τομεί. Στην Επιτροπή βεβαίως συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ένωσης και του Καναδά, εν προκειμένου στη ΣΕΤΑ γιατί τύπ θα είναι βέβαια Ένωση και Ενωμένων Πολιτειών. Τώρα, ε, αυτή οι joint Committee για ποια πράγματα μπορούν να λαμβάνουν δεσμευτικές αποφάσεις. Θα είναι τομείς ή είναι τομείς της ΕΤΑ που αναφέρονται ρητά μέσα στην συμφωνία. Λέει δηλαδή ότι στον τάδε ή τάδε πράγμα η Joint Committee μπορεί να λάβει δεσμευτική απόφαση. Έχω και ένα συνάδελφο που θεωρεί ότι οι τομείς αυτοί είναι τόσο ισχυροί που στην ουσία μειώνουν την κυριαρχία των χωρών μελών και τη Ένωση, κάτι το οποίο βέβαια θέτει θέμα δημοκρατίας. ποιο θα ελέγχει τα πράγματα αυτά, ποιο είναι αρμόδιος να κρίνει αν νομιμοποιείται δημοκρατικά. Μπορεί κανείς να το αποδυναμώσει κιόλα αυτό βέβαια και να εξετάσει τις ε, αρμοδιότητες αυτές λήψη αποφάσεων που συνήθω αναφέρονται σε κάποιε λεπτομέρειε βασικών κεφαλαίων. Δηλαδή, προβλέπεται, ας πούμε, προβλέπονται κάποιες εξαιρέσεις από τελωνιακούς δασμούς και μετά υπάρχουν ογλόγρα κατεβατά ε, λεπτομέρειες και πάνω εκεί αποφασίζει. Αυτό είναι και το σχήμα το οποίο προβλέπει τα διάφορα κεφάλαια και μπορεί να φανταστεί κανείς στην περίπτωση αυτή ότι για αυτά τα επιμέρους θέματα, έτσι είναι δηλαδή κιόλα, η μεικτή επιτροπή, η Joint Committee, μπορεί να λάβει δεσμευτικές αποφάσεις. Το ίδιο περίπου όπως οι εκτελεστικές πράξεις για ε, νομοθεσία που παράγει το Κοινοβούλιο. Μπορεί να πει κανεί ότι τέτοια πράγματα υπάρχουν και στις ε, ένομες χώρες, σε ένομες τάξεις των χωρών μελών και στην Ευρωπαϊκή. Το θέμα όμως είναι, και εδώ έγκυται η διαφορά σε αυτές τις διεθνείς συμβάσεις, ότι οι αποφάσεις αυτές δεν μπορούν πλέον να ανακληθούν. Αν δηλαδή ο Γερμανός υπουργό Συγκοινωνιών εκδώσει νέους κανόνες για τις μεταφορές στη Γερμανία, το Κοινοβούλιο μπορεί να βγει και να πει «Α, δεν μου αρέσουν, δεν συμφωνώ, για παράδειγμα αυτά τα πολύ μακριά φορτηγά, δεν μου αρέσουν, ανακαλώ την απόφαση αυτή». Τότε το διάταγμα του ε, Υπουργού Μεταφορών έχει ακυρωθεί. Αυτό το δικαίωμα ανάκρισης δεν υπάρχει βέβαια στην TTIP ή δεν θα υπάρχει. Εδώ βλέπω λοιπόν ένα σοβαρό πρόβλημα δημοκρατικής νομιμοποίησης το οποίο έχει συνέπειες και στις προδιαγραφές, τα στάνταρτ τα οποία είναι τέτοιες επιμέρους ρυθμίσεις όμως μπορεί να το αποφασίσει κανείς και συνολικότερα δηλαδή να πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Καναδική κυβέρνηση ή ενδεχομένως η Αμερικανική κυβέρνηση οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημο, ε, ε, νομιμοποιούνται δημοκρατικά με οποιοδήποτε τρόπο. Αν όμως αποφασίσει η καναδική κυβέρνηση, λείπει αυτή τότε η δημοκρατική νομοποίηση. Μου φαίνεται αυτό νομικά ε, σημαντικό. Δεύτερο τώρα, προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος και καταναλωτών. Στη διαπραγματευτική εντολή για την TTIP βεβαίως περιλαμβάνεται και το ότι επιθυμούμε να διατηρήσουμε υψηλά επίπεδα προστασίας ε, καταναλωτών και περιβάλλοντος. Βεβαίως. Αυτά μπορεί να μπουν και στο προήμιο της συμφωνίας. Αν όμως τα εξετάσει κανείς αυτά προσεκτικά, βλέπει και την παραπομπή στο περίφημο άρθρο 20 GATT, το οποίο πρέπει ωστόσο να ερμηνευτεί μόνο στη βάση του SPS, δηλαδή τη συμφωνία για φυτο-υγειονομικά μέτρα προστασίας και ούτω καθεξή και καταναλωτών κτλ. Δηλαδή πρέπει να το συναναγνώσει αυτό. Στις διαπραγματεύσει τώρα, και ελέγχθη αυτό προηγουμένω αντιπαρατάσσονται δύο νοοτροπίες, δύο φιλοσοφίες. Αφενό εμείς στην Ευρώπη έχουμε θεσπίσει και εθνικά και υπερεθνικά τη ρήτρα προφύλαξη που λέει ότι εάν κάτω από το επίπεδο κινδύνου. Υπάρχει έλλειψη γνώσης σχετικά με κάποιο στοιχείο το οποίο ενδέχεται να παράγει κίνδυνο, μπορώ να πω τότε προφυλακτικά ότι απαγορεύω την χρήση της ουσίας ή της τεχνολογίας ή ο καθεξής. Γενετική τεχνολογία, υδρορογμάτωση, άλλα σχετικά, τα οποία μπορεί κανείς να απαγορεύσει προληπτικά, προφυλακτικά. Οι Αμερικανοί τα γνωρίζετε αυτά, βεβαίως και από τις συζητήσεις για την προστασία του κλίματος κτλ. έχουν άλλη τοποθέτηση. Αυτοί θεωρούν ότι όσο δεν έχει αποδειχθεί ο συγκεκριμένος κίνδυνος επιστημονικά, είμαστε υποχρεωμένοι να επιτρέπουμε την χρήση των τεχνολογιών ή των μέσων. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι χειρότερο το σύστημα προστασίας του περιβάλλοντος που έχουν. Ξεκινά απλώς διαφορετικά, από διαφορετική αντίληψη. Έχουμε αποτελεσματικό δίκαιο προστασίας του καταναλωτού, ευθύνης δηλαδή του ρηπαίνοντο κλπ. Και αυτό επιβάλλουμε. Έρχεται επομένω εκ των υστέρων. Στι ευρωπαϊκέ χώρε δεν λειτουργεί καλά το σύστημα αυτό. Το εγχείρημα δεν προχώρησε, παρόλο που έγινε η προσπάθεια. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον στη Γερμανία, καμία απόφαση δικαστηρίου σχετική. Αν λοιπόν τώρα συνδυαστούν τα δύο συστήματα και πούμε ότι προχωρούμε τώρα προς μια εγκατάλειψη της αρχής της προφύλαξης και προχωρούμε προς την περιβαλλοντική ευθύνη, εκ των υστέρων δηλαδή, τότε μπορούμε να πούμε δεν με ενδιαφέρει αν πτωχεύσω διότι τα έχω βάλει τα λεφτά μου στην Ελβετία στο μεταξύ ή στο Λίχτενστάιν. Αυτή, είναι ο παραλληλισμός. Τώρα, τι, τι, σχέση έχει αυτό τώρα με τα φυτογειονομικά, SPS. Αυτά λένε ότι είναι εμπόδια στο εμπόριο και θα πρέπει να, περι, περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Αυτό όμως μόνο εφόσον έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι υπάρχει κίνδυνος από τα αγαθά αυτά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και το καθεξής. Η συμφωνία SPS, μάλλον στην συμφωνία SPS παραπέμπει η διαπραγματευτική εντολή TTIP και μάλιστα ρητά και η ΣΕΤΑ παραπέμπει ρητά στη συμφωνία SPS που λέει ότι η συμφωνία SPS συναποτελεί αναπόσπαστο μέρος και ισχύει απεριόριστα και μέσα στα πλαίσια της ΣΕΤΑ. Άρα βρισκόμαστε σε δυσκολίες με το, το σύστημα της προφύλαξης. Βεβαίω δεν πρέπει να ξαναγίνει το λάθος. Ο ΠΟΕ άλλωστε δεν λειτουργεί κατά τη γνώμη μου σωστά εδώ. Εάν όντως λειτουργήσει η ενδέχεται να οδηγηθούμε σε πολύ μοιραίες συνέπειες. Τρίτο σημείο, πάλι αναφέρεται στη δημοκρατία και στις προδιαγραφές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παραγάγει μια οδηγία η οποία θα οδηγούσε για τις παραχωρήσεις δηλαδή στην ιδιωτικοποίηση της παροχής νερού ξεκίνησε τότε ένα ευρύτατο ευρωπαϊκό κίνημα Right to Water με μια πετυχημένη πρωτοβουλία πολιτών και μάλιστα διπλά πετυχημένη διότι αφενός συνέλεξε τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών και δεύτερο είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ακυρώνουμε αυτό το εγχείρημα. Βέβαια δεν έχει πει την τελευταία της λέξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην ΣΕΤΑ ξαναβρίσκει κανείς ακριβώς αυτή την υποχρέωση διεθνών προσκλήσεων ενδιαφέροντος. Και πάλι μπαίνει το νερό εκεί. Και μάλιστα και παροχή νερού και αποχέτευση νερού. Άρα το ξαναβάζουν από το πίσω παραθυράκι, από την πίσω πόρτα. Αυτό αφορά αφενός στην δημοκρατική κήρυξη, δηλαδή κάποια στιγμή ξεκίνησε ένα δημοκρατικό κίνημα και είπε δεν τα θέλουμε αυτά τα πράγματα και τώρα με κάποιες αδιαφανείς διατάξεις πάει να πανέλθει. Το δεύτερο είναι ότι και βέβαια όταν γίνονται ε, δημόσιες προσκλήσεις εκδήλωση ενδιαφέροντος επιλέγονται οι πιο χαμηλές προσφορές. Οι χαμηλότερες προσφορές όμως δεν είναι απαραίτητο ότι σέβονται και τις διατάξεις προστασίας περιβάλλοντος και ούτω καθεξής. Και αυτό από την άποψη των προδιαγραφών που δεν είναι νομοθετικά ρυθμισμένες αλλά που έχουν θεσπίσει διάφορες αρχές, είτε σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτές ενδέχεται να υπονομεθούν και τελικά να τεθούν εκτός ισχύως. Ευχαριστώ. I thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Έρικ Γιόναρτ που είναι ο Γενικός ε, Γραμματέας της ε, Ευρωπαϊκής, ε, του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να σας δώσω μια μελέτη για το τι θα σημάνει ή θα μπορούσε να σημάνει η TTIP για την αυτοκινητοβιομηχανία. Ε, ε, θέλω λοιπόν εδώ να σας αναφέρω κάποια στοιχεία και νούμερα, διότι στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί φωνάζουμε όλοι για την TTIP, διότι είναι σημαντική όχι μόνο για τη δική μας βιομηχανία, αλλά και για τις θέσεις απασχόλησης. Άμεσα και έμεσα η αυτοκινητοβιομηχανία παρέχει απασχόληση σε 12,7 εκατομμύρια κόσμο. Ο τομέας μας στην Ευρώπη βασικά είναι εξαγωγικός τομέας. Παράγουμε περισσότερα από όσα πουλάμε εντός Ευρώπης. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι η TTIP είναι μια ευκαιρία να εξάγουμε ακόμα περισσότερα και άρα να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για απασχόληση εδώ στην Ευρώπη. Έχουμε αυτή τη στιγμή σαφείς φόρους, καθαρούς φόρους, ε, ε, από το εμπόριο 95,1 δις. Ε, ενώ όταν βλέπουμε τις εισαγωγές από ό,τι είπα στην Ευρώπη φτάνουμε περίπου στο 200.000 ε, ενώ εξάγουμε περισσότερα. Εξάγουμε περισσότερα από όσα εισάγουμε αυτοκίνητα. Στην TTIP έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας με τους ε, Αμερικανούς ε, εταίρους μας, ΑΣΕΑ, AAPC, ε, καθώς και την συνεργασία Alliance που αντιπροσωπεύουν την αυτοκινητοβιομηχανία των ΗΠΑ. Είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι στη θέση μας για αυτές τις διαπραγματεύσεις ελευθέρω εμπόριο. Ε, θέλουμε μια συνολική συμφωνία, όχι μόνο την κατάργηση των δασμών. Θεωρούμε πως πρόκειται για μια κολοσσία ευκαιρία ώστε να αντιμετωπίσουμε τα μη δασμολογικά, τους μη, δασμολογικούς φραγμούς ε, και την ε, νομοθετική ρύθμιση. Για μιας βέβαια, εφόσον βλέπουμε πόσο περίπλακο είναι αυτό, διακρίνουμε ανάμεσα στο τι μπορούμε να αναμένουμε σε σχέση με τις ισχύσεις νομοθεσίες ε, και τι να περιμένουμε από τη μελλοντική νομοθεσία. Για την, για την ισχύουσα νομοθεσία και αυτό ήδη αναφέρθηκε από την Κομισιόν όταν μίλησαν για ε, την αμοιβαία αναγνώριση αντιστοιχίας της νομοθεσίας μεταξύ Ένωσης και ΕΙΠΑ, ΕΕ, αλλά είμαστε και επιλεκτικοί Γνωρίζουμε δηλαδή ότι έχουμε τεράστιο έργο μπροστά μας, οπότε εστιάζουμε στις συζητήσει μας μόνο σε αντιστοιχεία νομοθεσίας περί ασφάλειας. Αν θέλαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, για κάθε νομοθεσία που ισχύει θα ήταν αδύνατη υποστολή. Άρα λοιπόν εστιάζουμε στην ασφάλεια και αυτό για τα επιβετικά αυτοκίνητα. Όταν πρόκειται για φορτηγά, εδώ δεν εισάγονται ούτε εξάγονται φορτηγά ολόκληρα, αλλά οι κινητήρες αυτών. Και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε στην ε, ανημιδέα αναγνώριση αντιστοιχίε ε, όσον αφορά τα πρότυπα εκπομπών ρήπων για τα εμπορικά αυτοκίνητα, τους εμπορικούς κινητήρες βασικά. Και εκεί θα θέλαμε στη μελλοντική μας νομοθεσία να προχωρήσουμε προς εναρμόνιση. Τώρα, κάποιος από τους προηγούμενους ομιλητές μίλησε για το πώς και τι εγώ θα ήθελα να μιλήσω για το πώς. Ποια είναι η διαφορά για το πώς ρυθμίζεται ο δικός μας ε, τομέας ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Ένωση. Τελικά, τελικά, στην Ευρώπη έχουμε, έχουμε μία ειδική έγκριση Μπορεί δηλαδή κανείς να εμπορευτεί αυτοκίνητα μόνο από τη στιγμή που έχουν εγκριθεί από την Εθνική Αρχή ότι είναι σύμμορφα προς ε, τη συγκεκριμένα στάνταρ και νομοθεσίες, ενώ στις είπα όταν εστιάσει κανείς στην ασφάλεια πρόκειται για ένα σύστημα αυτοπιστοποίησης. Ο κατασκευαστής δηλαδή πρέπει να πιστοποιήσει ότι συμμορφούνται προς τις αρχές, προς τις νομοθεσίες και τότε οι αρχές μπορούν να ελέγξουν κατά πόσο αυτό ή όχι Ε, δεν χρειάζεται λοιπόν να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτή είναι η δασική διαφορά. Τώρα, ποιες είναι αυτές οι νομοθεσίες. Αν δούμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ο τομέας μας ρυθμίζεται καταρχήν από τις παγκόσμιες τεχνικές προδιαγραφές, από την άλλη πλευρά από τις προδιαγραφές του ΟΗΕ και από τις προδιαγραφές της Ένωσης. Τρία σύνολα προδιαγραφών από τη ΣΥΠΑ έχουν παγκόσμιες τεχνικές ρυθμίσεις και από την άλλη πλευρά, όταν εστιάσουμε στην ασφάλεια, όπως είπαμε και πριν, έχουμε πρότυπα ασφαλείας αλλά και κανονισμούς που ορίζει η Νίτσα. Και πάλι εδώ έχουμε του κανονισμούς που ορίζει η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, WP29, 59 χώρε συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, αλλά εκεί δεν περιλαμβάνονται οι ΙΠΑ. Και, έχουν και ασχολούνται με έναν μεγάλο φάσμα προδιαγραφών, φωτισμός, περιβαλλοντικά, ζώνες ασφαλείας, ε, δοκιμές ε, για ατυχήματα, συγκρούσεις κτλ. Πρόκειται για ένα πολύ προηγμένο σύνολο κανονισμών του ΟΗΕ και είναι 108 αυτές οι ρυθμίσεις, οι προδιαγραφές που διέπουν το δικό μας τομέα. Μετά έχουμε ειδικέ διατάξεις της Ένωσης όσον αφορά τη γενική ασφάλεια, την προστασία των πεζών κτλ. διαστάσεις. Τώρα και στους δύο ε, ισχύουν αυτές οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές που υιοθετούνται στο πλαίσιο της Συμφωνίας του 98 για τις γενικές ε, παγκόσμιες τεχνικές προδιαγραφές του ΟΗΕ. Αυτά ισχύουν και από τις δύο πλευρέ και μετά στη ΣΥΠΑ υπάρχουν και οι προδιαγραφές του Νίτσα που είναι η ρυθμιστικός οργανισμός για τις μεταφορές και ε, λογοδοτεί στο Κογκρέσο. Όλα αυτά λοιπόν ισχύουν στο πλαίσιο της αυτοπιστοποίησης. Υπάρχουν διαφορές, ομολογουμένως, αλλά και τα δύο σύνολα των ρυθμιστικών προδιαγραφών προσφέρουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο απόδοσης όσον αφορά την ασφάλεια για τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ωστόσο, αυτές οι ρυθμιστικές διαφορές απαιτούν από τους κατασκευαστές να δημιουργήσουν διαφορετική δομή και σχεδιασμό για τα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ένωση ή τα οχήματα που κυκλοφορούν στις ΗΠΑ. Να πούμε διαφορετικό σασί, διαφορετικοί καθρέφτες, διαφορετική καφότα ε, προβολής. Διαφορές που ωστόσο δεν οδηγούν από, από, σε επιπλέον ασφάλεια και αυτό είναι και το συμπέρασμα των δικών μας μελών που, που δουλεύουν και από τις δύο όχθες του Ατλαντικού. Φυσικά το να ανταποκριθεί κανείς και στα δυο σύνολα προδιαγραφών κοστίζει πολύ. Κανένα από τα δύο συστήματα δεν είναι πιο ασφαλές, είναι απλώ διαφορετικά. Ξέρουμε ότι η εναρμόνιση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία θα είναι πρόκληση δεδομένου ότι οι ίδιοι κανονισμοί αυτοί είναι διαφορετικοί. Ο τομέας, μα το έχει ήδη προσπαθήσει αυτό παλιότερα, να προσπαθήσει δηλαδή να αρμονίσει τα αυτοκίνητα και απέτυχε κατά τη διάρκεια του διατλαντικού διαλόγου. Θα πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας λοιπόν και γι' αυτό βλέπουμε ότι η λύση για τις ισχύουσε νομοθεσίες, όχι για τις μελλοντικές αλλά για τις ισχύουσε είναι να προχωρήσουμε προς μια αντιστοιχία. Αναγνώριση και αντιστοιχία των κανονισμών. Είμαστε της άποψης λοιπόν ότι ο κανονισμός της Ένωσης και τον είπα για τα αυτοκίνητα, τα επιβατηγά επιτυγχάνουν την ίδια απόδοση όσον αφορά την ασφάλεια αυτό για τα επιβατικά αυτοκίνητα. Όσον αφορά τα εμπορικά οχήματα, χορτηγά, εκεί θέλουμε να έχουμε αντιστοιχεία για τις προδιαγραφές εκπομπών, το Euro 6 όπως λέγεται, ενώ στην Αμερική λέγεται EPA 10. Και πάλι, ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός με βάση τη Washington που παρέχει επιστημονικές αναλύσεις στους ε, ρυθμιστές της ε, περιβαλλοντικής, ε, των περιβαλλοντικών διδάξεων έκαναν σύγκριση ανάμεσα στα στάνταρ που ισχύουν στη ΣΥΠΑ και στην Ένωση και κατέληξαν ότι είναι αντίστοιχες επιλογές και απαιτούν τους ίδιους, ε, τις ίδιες τεχνολογίες ελέγχου ρήπων και επιτυχάνουν τα ίδια ωφέλη όσον αφορά τις εκπομπές ρήπων. Εμείς συλλέγουμε στοιχεία από τα μέλη μας ώστε όντω να επιβεβαιώσουμε πως ε, τα δύο σύνολα προδιαγραφών ε, έχουν παρόμοια απόδοση. Τώρα, πώς συμβάλλουμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Εμείς ε, στηρίζουμε τη διαπραγματεύση. Είναι περίπλοκη, περίπλοκο το θέμα και γι' αυτό και συμφωνήσαμε να κάνουμε μελέτες και κάθε φορά που γίνονται συνεδριάσεις των ε, εμπλεκόμενων φορέων να ενημερώνουμε όχι μόνο την Κομισιόν αλλά και τους, ε, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Και αυτή τη στιγμή γίνονται δύο μελέτες που είναι υπό εξέλιξη. Μία είναι τεχνικής φύσης που γίνεται από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν στις ΗΠΑ και από το Πανεπιστήμιο του Τσάρμες στην Σουηδία και προσπαθούν να αποδείξουν την αντιστοιχεία των ενωτικών και των αμερικανικών προδιαγραφών για τα επιβατικά αυτοκίνητα όσον αφορά την ασφάλεια. Με πρόσβαση στα στοιχεία που υπάρχουν στις δυο επίρου είμαστε στην τελευταία φάση της μελέτης και τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα σύντομα. Έπειτα, επειδή συχνά παίρνουμε ερωτήσει για το τι σημαίνει όλο αυτό από οικονομικής άποψης, εμείς συνεργαζόμαστε με την έρευνα ε, της αυτοκινητοβιομηχανίας για να δείξουμε ποια είναι τα συμφέροντα, τι έχουμε να κερδίσουμε από τη ρυθμιστική σύγκληση στην TTIP. Πάντως, σαφώς, οι μεγαλύτερε ευκαιρίε είναι στην ρυθμιστική σύγκληση. Αν δεν εξετάσουμε τι διαφορέ κανονισμών σήμερα, δηλαδή μη δεσμολογική φραγμή στι δύο περιοχέ αυτού του κόσμου, ε, αποτιμώνται από το Κέντρο Ερευνών Οικονομικής Πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου ότι αντιστοιχούν σε έναν δασμό περίπου 26%. Εάν δηλαδή μπορούσαμε αυτό να το καταργήσουμε, θα έχουμε πολύ μεγάλες εξοικονομήσεις κόστου κατάργηση των δασμών για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές, καθώς και 25% των υφιστάμενων NTB, μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση των εξαγών προς τη ΣΥΠΑ κατά πάνω από 100% υπολογίζουμε. Και πάλι, Εξοικονομήσει από του δασμού είναι σημαντικέ, αλλά τα μεγαλύτερα ωφέλη θα προέκυπταν από την ρυθμιστική σύγκληση και γι' αυτό και επιδιώκουμε μια συνολική καθολική συμφωνία που θα περιλάμβανε και τη ρυθμιστική σύγκληση. Και έρχομαι στα συμπεράσματά μου κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει λοιπόν όντως να καταργηθούν τα ρυθμιστικά, οι ρυθμιστικοί φραγμοί για τις ισχύουσες νομοθεσίες εδώ δεν θέλουμε να μειώσουμε τις προδιαγραφές μας, όχι. Θέλουμε να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση και αντιστοιχεία των ισχυών των, ισχυών των ε, κανονισμών ασφαλής και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε. Να γνωρίζετε δε ότι το εμπόριο των αυτοκινήτων αντιπροσωπεύει το 10% του συνολικού εμπαρίου μεταξύ ε, ε και είπα. Άρα το δυναμικό για τις οικονομίες στις δύο περιοχές του κόσμου αυτού, αυτές θα είναι απίστευτο. Θα αυξήσει το ρόλο το... της Ένωσης αλλά και των ΙΠΑ ως ε, παγκόσμιων υποδειγμάτων στις προδιαγραφές. Είναι ευκαιρία για την Ευρώπη για θέσεις απασχόληση, ανάπτυξη και σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία να σας δώσουμε τη δική μας προοπτική και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για ερωταπαντήσεις. Ε, σας ευχαριστούμε τα μάλα και τώρα τα ερωτήματα των μελών και η πρώτη είναι η κυρία Κέλλερ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ομιλητές. Δεν έχω τόσο πολλές ερωτήσεις. Απλώς θα ήθελα η να αντιδράσει σε αυτά που είπαν οι ομιλητές σε σχέση με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και είπατε πολλά πράγματα τα οποία δεν αντιμετωπίζει το Συμβούλιο Ρυθμιστικής Συνεργασίας. Γιατί αυτό που είπατε ότι κάνει είναι προωθεί την εναρμόνιση κτλ. Όλα αυτά δεν είναι δράση. Αυτά είναι στοχοθεσία. Ποιε είναι οι δράσει, ποιε είναι οι αρμοδιότητε του Συμβουλίου Ρυθμιστική Συνεργασία και τι θέλετε να πείτε απαντώντας για τις λεγόμενες ζωντανές συμφωνίες. Τι σημαίνει αυτό. Έχετε μια συμφωνία που ακόμα δεν έχει το περιεχόμενό της και το οποίο θα προσθεθεί αργότερα. Είπε η Κομισιόν ότι τα περισσότερα ε, ωφέλη σε οικονομικό επίπεδο θα έρθουν από αυτή τη ρυθμιστική συνεργασία. Πώς εξασφαλίζετε λοιπόν ότι θα γίνει κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα. Ο κύριος Σιόλτς. Σας ευχαριστώ και εγώ έχω ένα ερώτημα προς την Κομισιόν. Συγκεκριμένο ερώτημα. Ξέρουμε ότι με αυτή τη συνεργασία σε ρυθμιστικό επίπεδο θα υπάρχει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Θα υπάρχει λοιπόν μια δυνατότητα έγκαιρης συνεννόησης για ορισμένα ρυθμιστικά συστήματα, ε, ε, ρυθμιστικά ερωτήματα. Αλλά ένα τέτοιο ερώτημα ε, συνδέεται με το ποιος θα κάνει την τελική εκπόνηση των κανόνων. Θα εμπλέκονται οι επενδυτές στην διαδικασία αυτή για την εκπόνηση ρυθμιστικών κανόνων ή θα εμπλέκονται οι κοινοβουλευτικοί την ε, ρύθμιση των μελλοντικών κανόνων. Αυτοί που εκπροσωπούν το δημόσιο συμφέρον δηλαδή. Ο κύριος Λεμπρετό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από όλα θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή Ανδρέας Φιζάν για την λαμπρή του παρέμβαση που επιβεβαιώνει τις δικές μου αναλύσεις για το πόσο επικίνδυνη είναι η ΣΕΤΑ και η TTIP προς τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, ο οποίος προσπάθησε να μας διαβεβαιώσει για την εναρμόνιση των ρυθμίσεων. Μας, μας εξήγησε ότι η TTIP δεν είναι τόσο επικίνδυνη, ότι είναι λίγοι οι τομείς οι οποίοι θα καλυφθούν και μας έδωσε ένα παράδειγμα εναρμόνισης, ένα παράδειγμα το οποίο το ανέφερε και ένας άλλος ο μιλητή που είναι η αυτοκίνητο βιομηχανία. Το πρώτο ερώτημα είναι, μπορεί να μα δώσει κάποιον άλλο τομέα ο οποίο απετέλεσε αντικείμενο εναρμόνιση μέσα στην TTIP και δεύτερο, το θέμα των προελεύσεων, ε, των ονομασιών προέλευση που προστατεύονται. Εδώ η Κομισιόν θα πρέπει να διαπραγματευτεί για τα θέματα αυτά μέσα στην TTIP. Μπορεί να μας διαβεβαιώσει ο πρόσωπος TTIP ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τις ορμασίες προέλευσης που προστατεύονται θα διατηρηθούν, ναι ή ου. Κύριος Φως. Ευχαριστώ πολύ. Ερώτηση προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κύριο Πίνινγκ και μετά στον κύριο Φίζαν. Πίνινγκ. Διάβασα σε μια μεγάλη γερμανική εφημερίδα σήμερα ότι θα δοθεί στους Αμερικανούς κάποιο δικαίωμα συμμετοχής ή τέλο πάντων να έχουν λόγο στην ε, νομοθετική διαδικασία. Ε, γιατί είναι σωστή είδηση αυτή. Πού βρίσκονται τα πράγματα. Φύζαν δύο πράγματα που δεν κατανόησα πολύ καλά. Αναφέρατε παραπομπή στον ΠΟΕ και στην ΚΑΤ που τα κρίνεται πολύ αρνητικά. Αλλά πόσο ξέρω είναι ισχύον δίκαιο και που εφαρμόζεται μάλιστα εν μέρη και στις χώρες μέλη μας. Έτσι λοιπόν, εγώ δεν το βλέπω τόσο αρνητικά. Σε ό,τι αφορά ε, τα όσα είπατε για το νερό, ως παράδειγμα, και ως σκανδαλώδες, αυτό είναι σωστό μόνο όπου η τοπική κοινότητα έχει αποφασίσει να ιδιωτικοποιήσει όντως την παροχή νερού. Και τότε μόνο γίνονται προσκλήσει εκδήλωση ενδιαφέροντος. Όχι όμως εάν η τοπική κοινότητα δεν αποφασίσει να ε, ιδιωτικοποιήσει την παροχή νερού και συνεχίζει να το έχει στην δική της ε, διαχείριση. Ευχαριστώ. Εσείς, κυρία Κέλλερ. Ναι. Όπως ο κύριος Βόσο, διάβασα και εγώ το σχετικό άρθρο που λέει ή παραθέτει τέλο πάντων ότι και από κεντρωμένα επίπεδα θα συμμετέχουν και θα παρέχουν προφορίες τα Ε, τι είναι αυτό, τι είναι αυτά τα αποκεντρωμένα επίπεδα, περιφερειακές διοικήσεις. Δεν φτάνω να διαβάσω το όνομά σας κύριε μου, κάντε μια σύντομη ερώτηση. Α, Ροδρίγης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. χρειάστηκε να απουσιάσω και έχασε ένα κομμάτι της συζήτηση, που είναι εξαιρετικά σημαντική και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και επικοδομητική. Ήθελα να κάνω μια σκέψη και επίση να, να αναφερθώ σε δύο ερωτήματα. Η σκέψη μου είναι η εξή. Ένα από τα κύρια προβλήματα τα οποία επηρεάζουν το εμπόριο και την ισότητα ανταγωνισμού είναι ακριβώς τα μη, η μη ε, τελωνιακή φραγμή η ρυθμιστική φραγμή, η τεχνική και διοικητική φραγμή κτλ. Είχαμε την ευκαιρία, πιστεύω, πολλοί από τις βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή ΙΝΤΑ να γνωρίσουμε την πραγματικότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλές από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στο διεθνές εμπόριο. Υπάρχει μια μεγάλη προσδοκία ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό και να ξεπεράσουμε τα αριθμιστικά εμπόδια, να υπάρχει μεγαλύτερη εναρμόνιση. Το ερώτημά μου είναι κατά πόσο θα καταστεί σύμφωνο, καταστεί δυνατό να ανταποκριθούμε στις ε, προσδοκίες αυτές με την TTIP ή αντίθετα θα δημιουργηθεί μια ματέωση σε αυτό το κέριο τομέα. Το άλλο ερώτημα το οποίο ήθελα να θέσω είναι πώς βλέπετε την προοπτική της ρύθμισης για τα εργασιακά δικαιώματα μέσα στην TTIP, σε ποιο βαθμό θα καταστεί δυνατό, αν είναι δυνατόν, να υπάρξει μια συμφωνία που θα εμποδίσει να ισοπεδωθούν προς τα κάτω τα πρότυπα και επίσης αν είναι εφικτό να εξασφαλίσουμε ότι στο μέλλον μέσα από τη ρυθμιστική ε, ε συνεννόηση να υπάρξουν νέες συμφωνίες για τα εργασιακά. Και τώρα οι ίδιοι ακεκριμένοι ομιλητές μας έχουν την ευκαιρία να λάβουν το λόγο για 1,5 λεπτό καταρχήν, αλλά όχι. Αστείευομαι όσο πιο σύντομα μπορείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φοβάμαι ότι η ποιότητα της απάντησης θα εξαρτηθεί από το χρόνο που είναι διαθέσιμος. Μπορώ να σας πω κάποιες γενικότητες, αν οι γενικότητες ε, λυπάμαι, θα μπορώ να επεκταθώ περισσότερο αν με αφήσετε. Τι θα έκανε ένα σώμα Ρυθμιστική συνεργασία. Πρώτον, να παρακολουθεί την εφαρμογή των ρητρών, να εποπτεύει το ρόλο των ρυθμιστών και να εγκρίνει σχέδια ώστε οι ρυθμιστές και από τις δύο πλευρές να δούνε πού ακριβώς θα πρέπει να συνεργαστούν στο μέλλον. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να εντοπίσουν ευκαιρίες για να υπάρχουν νέοι κανόνες ή να υπάρξει μεγαλύτερη συμβατότητα των κανόνων. Αυτό είναι ο κύριος στόχος του Συμβουλίου. Οποιοςδήποτε λοιπόν που θέλει να θέσει ένα θέμα ρυθμιστικού χαρακτήρα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να φτάσει σε ένα φόρουμ, είναι ένα συμβουλευτικό φόρουμ, το συμβουλευτό δεν παίρνει αποφάσεις. Μια ζωντανή συμφωνία, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να περατώσουμε όλα αυτά που θέλουμε να πετύχουμε στους διάφορους τομείς, θα υπάρξουν περαιτέρω πρόνοιες που θα πρέπει να γίνουν στο μέλλον και θα πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε αυτή η νέα συνεργασία να αντανακλάται σε πρόνοιες που θα εφαρμοστούν αργότερα. Δεν ξέρουμε πώς θα γίνει προς το παρόν. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει κάτι τέτοιο. Πάντως προτού υπάρξει νέα, νέες ρήτρες συνεργασίας θα πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες διαδικασίες διαβούλευσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ε, διαβούλευση με τα νομοθετικά σώματα τα οποία είναι αρμόδια. Δεν υπάρχει περίπτωση ένα σκοτεινό όργανο να πάρει αποφάσεις για θέματα που αφορούν τους Ευρωπαίους πολίτες. Σε ό,τι αφορά τα παραδείγματα. Σε άλλους τομείς, φαρμακευτικός τομέας. Μπορεί να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση επιθεωρήσεων, εγκαταστάσεων, παρασκευής ε, φαρμάκων και ιατρικών συσκευών. Και έτσι δεν θα χρειάζεται να υπάρχει διπλή επιθεώρηση. Θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερη σύγκριση στα κριτήρια και τις διαδικασίες τεχνικής Αξιολόγηση ουσιαών και σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να υπάρξει ανταλλαγή δεδομένων και μπορεί να υπάρξει μικρότερη έτσι ανάγκη για να παρουσιάζουν οι εταιρείε δύο διαφορετικούς φακέλους σε εθνιστικές αρχές. Αυτά. Επίσης για την ονομασία προέλευσης δεν υπάρχει καμία ιδέα να αλλάξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση το καθεστώς της. δεν θα υπάρξει δυνατότητα λήψης απόφασης από κανένα σώμα εάν δεν μπορούν να συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές για οποιοδήποτε το οποίο θα έχει άμεση εφαρμογή. Δεν θα υπάρχουν νέοι κανόνες οι οποίοι θα προκύψουν από οποιοδήποτε φορέα της Τσιτσίπ. Πιστεύω λοιπόν ότι για αυτόν ακριβώς τον λόγο όλα αυτά τα οποία θα αποφασιστούν στην TTIP θα πρέπει να υπόκειται στον απαραίτητο δημοκρατικό έλεγχο δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατικό έλλειμμα. Και όταν πρόκειται για τους κανόνες του ΠΟΕ και τα φυτοϊγειονομικά μέτρα, δεν χρειαζόμαστε την TTIP για να εφαρμόζονται οι αρχές αυτές παντού. <clears throat> Ο ΠΟΕ ήδη επιβάλλει τέτοιου είδους υποχρεώσεις για τις κοινοφελείς επιχείρησεις όπως αναφέρθηκε προηγουμένως από κάποιον ομιλητή Μιλάμε για τομείς όπου υπάρχει ήδη ανοιχτός χαρακτήρας σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αναλάβει δεσμεύσει για τις ανοιχτές διαδικασίες προμηθειών. Δεν υπάρχει τίποτα καινούριο λοιπόν και εμείς θα το διατηρήσουμε αυτό, θα διατηρήσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες. Και οι πράξεις οι οποίες δεν είναι σε κεντρικό επίπεδο, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι συζήτηση αλλά <clears throat> κατά πάσα πιθανότητα η αρχική μας πρόταση θα είναι να εστιάσουμε στην, ε, στις πράξεις σε κεντρικό και ομοσπονδιακό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να φτάσουμε σε λεπτομερείς υποχρεώσεις για διαφάνεια και διαβούλευση, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι υπό ε, Τέλος, θα μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες. Είναι τεράστιες οι προκλήσεις, για να μην Ξέρουμε πόσο δύσκολο ήταν να έχουμε μία ενιαία αγορά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την μια πλευρά θα πρέπει να έχουμε υψηλέ φιλοδοξίε, αλλά από την άλλη πλευρά ξέρουμε ότι θα χρειαστεί χρόνο για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το οικοδόμημα. Τα εργασιακά δικαιώματα δεν θα φυγούν, δεν είναι υποσυζήτηση και η συμφωνία θα περιέχει επίσης μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης για να εμποδίσει τη δημιουργία νέων φραγμών ώστε όταν οι ρυθμιστές σκέφτονται τους νέους κανονισμούς, η άλλη πλευρά θα ξέρει εάν υπάρχει κάτι δυνητικά εμποδιακού χαρακτήρα και θα υπάρξει μια ανταλλαγή απόψε μεταξύ τους. Thank Σας ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Από τους άλλους κυρίως, κανείς επιθυμεί να λάβει το λόγο για να απαντήσει. Ναι, σύντομα, πρώτη ερώτηση του κυρίου Βος για το εάν οι Ενωμένε Πολιτείε θα παίξουν κάποιο ρόλο στην νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε μαζί με τους stakeholder να ε, έχει φωνή στις ε, νομοθετικές διαδικασίες στις Ενωμένες Πολιτείες και οι δύο πλευρές. Στην TTIP βεβαίως δίνουμε τυπική μορφή στη διαδικασία αυτή. Και έρχομαι και στην πρώτη ερώτηση της κυρίας Κέλλερ που ρώτησε πού εντοπίζεται η δράση. Μπορεί το Ρυθμιστικό Συμβούλιο να προωθήσει κάποιες ενέργειες. Όχι, είπατε, σας είπαν ότι θα είναι μάλλον όργανο που θα παρακολουθεί. Άρα, για τη νέα νομοθεσία όπου θα υπάρχει ένα εγγενές σύστημα, ένα είδος δηλαδή υποχρέωσης και των δύο ρυθμιστών για να συνδιαλέγονται όταν θα υπάρχει χώρος για κοινέ ρυθμίσεις. Άρα θα λέει η βιομηχανία ας αρχίσουμε να συζητούμε αν έχουμε κοινά δεδομένα και να αρχίσουμε την νομοθετική διαδικασία μετά, να την προωθήσουμε δηλαδή στο Κοινοβούλιο. Ε, professor Fizan; Εσείς κύριε καθηγητά Φιζάν. Ναι, τρεις ερωτήσεις. Πρώτη, δεν προϋποθέτουν οι ε, προσκλήσεις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος ότι έχει ιδιωτικοποιηθεί η απόφαση, υπάρχει απόφαση για ιδιωτικοποίηση της ε, παροχής νερού. Όχι απαραίτητα, μπορούν να είναι και άλλοι φορείς. Μπορούν να είναι δηλαδή και τυπικά ιδιωτικοποιημένες μορφές ε, εργασίας των Δήμων. Δεύτερο, υπάρχει και συμφωνία SPS, όπου είναι ακόμα εν και εφόσον παράγουμε νέα νομοθεσία θα πρέπει να συζητούμε και το χειρότερο ενδεχόμενο σενάριο. Και εκεί η TTIP μπαίνει στο παιχνίδι. Τα γνωρίζουμε δηλαδή και από το ευρωπαϊκό δίκαιο ότι υπάρχουν διατάξεις που και μετά από μία τριακονταετία ξαφνικά καθίστανται ενεργές. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με το dispute settlement. Και αυτό το χειρότερο σενάριο δηλαδή είναι που ενδιαφέρει τους νομικούς. Τρίτο, τι γίνεται με την εναρμόνιση δεσμευτικά, δεσμευτικές ε, δικαιωτικέ ρυθμίσει κτλ. Τα λέει αυτά ο κ. Όσο λειτουργούν τα κοινοβούλια και αποφασίζουν κατά αρμοδιότητα, καθαρά νομικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί οι προτάσει μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Μετά όμω μπαίνει πολιτικά το ερώτημα ποιε στην πράξη δεσμεύσει υπάρχουν. Πώ μπορεί δηλαδή να επιφέρει μικρές διορθώσει το Κοινοβούλιο σε κάποιες αποφάσεις που έχει ήδη λάβει η Joint Committee. Αυτό όμως είναι, είναι ξεκάθαρο, είναι ξεχωριστό μάλλον από το αν νομιμοποιείται δημοκρατικά. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Κύριε Ζωνάτ. Καθώς προχωράμε προς το τέλος της ε, συνεδρίας, όχι ευχαριστώ πρόεδρε. Uh, thank you. Ε, Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Τώρα. για το τελευταίες παρατηρήσεις θα ήθελα ο κύριος Άλεξ Φως να πάρει το λόγο γιατί είναι ο συντάκτης ε, για λογαριασμό της ε, Επιτροπής Ζούρη για τη γνωμοδότηση περί, σχέσεων, περί της έκθεσης ε, των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις τη, για την TTIP. Θα προσπαθήσω, ευχαριστώ πολύ, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Αφενός, οφείλω να πει κανείς ότι η ISDS βέβαια αμφισβητείται πολύ, είναι πολύ αμφιλεγόμενη στην κοινή γνώμη. Όμω, άκουσα εδώ τη συζήτηση ότι πρώτον είναι απαραίτητη, είναι αναγκαία η προστασία των επενδυτών. Άλλωστε στι διεθνεί οικονομικές σχέσεις είναι κατεστημένο όργανο αυτό. Ανταποκρίνεται στα, στα ευρωπαϊκά συμφέροντα και υποτίθεται ότι μειώνει ή αποκλεί οποιασδήποτε αυθαιρεσίες. Για μένα λοιπόν είναι καθαρό ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα ορισμένο πώς προστατεύονται οι επενδυτές, πώς λειτουργούν τα διαιτητικά δικαστήρια. Ακούσαμε άλλωστε τι γίνεται με τις εναλλακτικέ επιλογές, εδώ ίσως συνοπτικά βέβαια, αλλά και ποια είναι η πρακτική εφαρμογή για την αντιμετώπιση διαφόρων άλλων προβλημάτων ή μάλλον ότι αυτή έχει και άλλα προβλήματα και ενδεχομένως δεν ανταποκρίνεται πάντοτε στις ανάγκες, τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα. Και ότι το μέχρι τώρα ε, ισχύον μοντέλο θα πρέπει να γίνει πιο επίκαιρο και να προσαρμοστεί, να εξυγχρονιστεί. Ακούσαμε και διάφορες άλλες προτάσεις για διαιτησία, για εφέσεις, δηλαδή ε, επίπεδο εφέσεων και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι συνολικά ένα βασικό, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι έχει έρθει πλέον η ώρα το σύστημα ISDS να βασίζεται σε διαφανείς δομές, όποια και αν είναι η μορφή που θα λάβουν εν τέλει, χρειάζεται ωστόσο κάποια δομή και χρειάζεται μάλιστα και μια περαιτέρω εξέλιξη της δομής αυτής και εν τέλει τα διευθυντικά δικαστήρια φαίνεται να είναι αναγκαία ή τουλάχιστον να είναι μια οδός για την επίλυση των διαφορών. Πάντως δεν φαίνεται να ανοίγεται η οδός να μην, διπλή αντική διατύπωση δηλαδή, να μην προβλεφθεί απολύτως καμία διαιτητική διαδικασία. Νομίζω ότι πρέπει να τονίσω και πάλι την ανάγκη να υπάρξει μια δομή, γιατί αυτή ανοίγει βέβαια και την διαφάνεια. Επιτρέπει δηλαδή να υπάρξει διαφάνεια εφόσον υπάρχει δομή. Ε, thank Ευχαριστώ κύριε Φως. Έξω ονόματος των δύο επιτροπών και των προέδρων τους ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διακεκριμένους καλεσμένους και ομιλητές μας για τις παρουσιάσεις τους και όλους σας για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ.